Καλημέρα σας αγαπητοί συνάδελφοι. Παρακαλώ καθίστε για να ξεκινήσουμε με το σημείο 15 την παρουσίαση από την Προεδρία του Συμβουλίου την Europol και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη σύνδεση της Δανίας με την Europol μετά την 1η Μαΐου 2017. Όπως ξέρετε, μετά το δανέζικο δημοψήφισμα, η κυβέρνηση της Δανίας ε, αναζητεί τρόπους για να συνεχίσει τη σύνδεσή της με τη Europol και μετά την 1η Μαΐου 2017 που θα τεθεί σε εφαρμογή ο νέος κανονισμός της Europol. Ξέρω ότι είστε εξοικειωμένοι με το θέμα οι παρόντες. Θα ήθελα πάντως να υπενθυμίσω σε όσους δεν το γνωρίζουν ότι έχουμε ξανασυζητήσει αυτό το θέμα στην Επιτροπή και μάλιστα θέσαμε, ε, δώσαμε τη θετική μας γνώμη για τη συμπερίληψη της Δανίας στον κατάλογο των τρίτων χωρών με τις οποίες η Ευρωπόλ δύναται να διαπραγματευτεί ε, συμφωνίες συνεργασίας. Και σήμερα το σχέδιο μιας τέτοιας ε, συμφωνίας επιχειρησιακής συνεργασίας θα μας ε, το παρουσιάσει πρώτα πρόσωπο τη Προεδρία του Συμβουλίου, κατόπιν εκπρόσωπο Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ένα εκπρόσωπο τη Europol. Θα ακολουθήσει η συζήτηση μετά την παρουσίαση και του δικού μας εισηγητή, του κ. Δίας Δεμέρα. Θα δώσω πρώτα το λόγο στον εκπρόσωπο της Προεδρίας, τον κύριο Τσιλιμπέρτη. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμη Ευρωβουλευτέ, θα κάνω μια σύντομη παρουσίαση, την οποία θα χωρίσω σε δύο τμήματα. Πρώτα θα εξάρω τον σημαντικό ρόλο που έπαιξε η Δανία στην εσωτερική ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδιαίτερα στη Europol και κατόπιν στο δεύτερο τμήμα θα σας παρουσιάσω τη διαδικασία που θα ακολουθήσουμε μετά την εντολή της 22ης Μαρτίου. Η παρούσα συνεργασία Δανίας-Europol είναι πολύ αποτελεσματική. Η Δανία είναι από τους ε, βασικούς ε, συμμετοχούς και χρήστες της ε, βάσης δεδομένων της Europol. Από, τις, από τα 29 εστιακά σημεία της Europol, η Δανία συμμετέχει ενεργά σε 25 τέτοια. Σε ό,τι αφορά και το σύστημα μηνύματος, ε, μηνυμάτων, η Δανία πρωτοστατεί σε ό,τι αφορά το σύγχρονο σύστημά της και σε ό,τι αφορά το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφοριών, το EIS, και εκεί η Δανία συμβάλλει με πο, πολύ αριθμ, μεγάλο αριθμό αναζητήσεων. Είναι η έβδομη σε ό,τι αφορά τις αναζητήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση από την Ευρωπαϊκή Βάση Πληροφοριών. Οπότε είναι σημαντικό να διασφαλίσουμε καλό επίπεδο συνεργασίας και μετά την 1η Μαΐου του 2017. Στόχος είναι να ε, περιορίσουμε στο ελάχιστο πιθανά κενά. Είναι γνωστή η διαδικασία που οδήγησε στη σημερινή ακρόαση. Όπως είπε και ο Πρόεδρος, το Συμβούλιο ζήτησε τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και το Φεβρουάριο το Συμβούλιο υιοθέτησε μία εφαρμοστική απόφαση που πρόσθεσε και τη Δανία στον κατάλογο των τρίτων χωρών. Άρα η Ευρωπόλ μπορεί να συνάψει συμφωνία με τη Δανία. Μάλιστα έχουν ξεκινήσει έκτοτε διαπραγματεύσεις και την περασμένη εβδομάδα το σχέδιο συμφωνίας επιχειρησιακής συνεργασίας ε, μεταξύ Δανίας και Γεωροπόλ απεστάλλει στο Συμβούλιο. Και κατόπιν στις 21 Μαρτίου υπευλήθηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η συμφωνία αυτή περιλαμβάνει και κάποια νέα στοιχεία σε σχέση με τις συνήθεις συμφωνίες ε, Europol και τριτοχωρών, χωρών, δεδομένης της δημοσιονομικής ε, κατάστασης ε, της Δανίας, που είναι και μέρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Σέγγεν. Πάντως, τις λεπτομέρειες της συμφωνίας θα μας παρουσιάσουν οι εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Europol μετά τη δική μου εισαγωγή. Αυτό που έχετε λάβει είναι το σχέδιο απόφασης επιχειρησιακής συνεργασίας που ε, χαράζει το δρόμο για την τελική υπογραφή της συμφωνίας αυτής πριν την 1η Μαΐου και θα ήθελα να τονίσω και κάτι πριν ολοκληρώσω, όπως ακούσαμε, ο μόνος τρόπος για να συμμετέχει πλήρως η Δανία στο νέο κανονισμό της Europol είναι να αξιοποιήσει τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 22 της Συνθήκων. Οπότε η σύναψη μιας συμφωνίας επιχειρησιακής συνεργασίας με τη Δανία δεν δυνατότητα πρόκειται να καταστήσει την Δανία μέλος της Europol. Απλώς εξασφαλίζει τη δυνατότητα μελλοντική συνεργασίας μεταξύ Δανίας και Europol, όπως ε, συμβαίνει και με άλλες τρίτες χώρες. Δεν δίνουμε όμως στη Δανία ε, μεγαλύτερη πρόσβαση ε, στη βάση των δεδομένων ή δικαίωμα συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων στην διακυβέρνηση της Europol. Αυτά και σας ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δώσετε να σας παρουσιάσω το σχέδιο της εφαρμοστικής απόφασης του Συμβουλίου και να υπενθυμίσω ότι δεδομένη του επίγοντος χαρακτήρα της σύναψης της συμφωνίας με τη Δανία και την Κυροπόλ θέλουμε να παρακαλούμε το Κοινοβούλιο να δώσει ιδιαίτερη προτεραιότητα και να διεκπαιρεώσει γρήγορα αυτή τη διαδικασία. Ευχαριστώ τώρα εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η κυρία Μίτσι. Ευχαριστώ και καλημέρα σας. Σήμερα ε, σημειώνεται ένα σημαντικό βήμα στη διαδικασία που το οδηγήσει στην ολοκλήρωση των διευθετήσεων που σκοπεύουν να επιτρέψουν να ελαχιστοποιηθούν ε, οι αρνητικές επιπτώσεις της αποχώρησης της Δανίας από το Europol. Το σχέδιο συμφωνίας, επί το οποίο το Ευρωπαϊκό, Κοινοβουλίο, ε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να εκφράσει την άποψή του, είναι παράρτημα ενός νομικού κειμένου που οι κύριοι Γιούνκερ Τούσκ και ο Πρωθυπουργό τη Δανία ε, σύνυψαν στι 15 Δεκεμβρίου. Το σχέδιο κειμένου αυτού επίση λαμβάνει υπόψη τι απόψει που εξέφρασε το Διοικητικό Συμβούλιο της Europol και τα μέλη του και τη γνώμη του Κοινού Υποπτικού Συμβουλίου της Europol καθώς και τη γνώμη που εξέφρασε το Κοινοβούλιο για την απόφαση να προσθεθεί η Δανία στο κατάλογο τρίτων χωρών με τις οποίες η Europol μπορεί να συνάπτει συμφωνίες. Τα μέτρα που προβλέπονται σε αυτή την κοινή δήλωση που προανέφερα αναφέρουν ε, ορισμένες σημαντικές ε, προϋποθέσεις οι οποίες είναι οι εξής. Πρώτον, η Δανία θα πρέπει να συνεχίσει να είναι μέλος της Ένωσης ε, και του χώρου Σέγγεν. Δεύτερον, η Δανία έχει την υποχρέωση να εφαρμόσει πλήρως στο εθνικό της δίκαιο την οδηγία για την προστασία των δεδομένων σε σχέση με τα αστυνομικά 6815 Και αυτή η εφαρμογή πρέπει να ολοκληρωθεί και να αρχίσει να ισχύει μέχρι την 1η Μαΐου τρέχοντος. Τρίτον, η Δανία πρέπει να συμφωνήσει ε, να επεκταθεί στο έδαφο της, στο έδαφος της η δικαιοδοσία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και του Ευρωπαϊκού Επόπτη Προστασίας Δεδομένων. Το σχέδιο κειμένου περιλαμβάνει αυτές τις προϋποθέσεις και να πω λίγα λόγια για να σας εξηγήσω γιατί αυτές οι προϋποθέσεις περιλαμβάνονται και πώς στο σχέδιο συμφωνίας. Ο ρόλος ε, του επόπτη προστασίας των δεδομένων, το 14C, αναφέρεται σε όλες τις σχετικές διατάξεις για την προστασία των δεδομένων που περιλαμβάνονται στο κανονισμό Europol. Η Δανία λοιπόν και η Europol δεσμεύονται κατά τις σχέσεις τους από τις διατάξεις του κανονισμού Europol που καθορίζει τις εγγύσεις για προστασία των δεδομένων που αποτελούν τμήμα του κανονισμού. Μεταξύ των οποίων αναφέρεται ο ρόλος του επόπτη προστασία δεδομένων όπως ακριβώς υιοθετήθηκε και από την Europol. Μόνο μία πλευρά επί της οποίας η θέση της Δανίας διαφοροποιείται από τα άλλα κράτη-μέλη. Λέγεται δηλαδή ότι η Δανία δεν συμμετέχει στο Συμβούλιο Συνεργασίας. Κατά τα άλλα συμμετέχει ισότιμα. Όπως επίσης είπα, το άρθρο 14D τονίζει ότι από την 1η 5η 17 η Δανία θα εφαρμόσει τους κανόνες που περιλαμβάνονται για την προστασία των δεδομένων για αστυνομικά θέματα στη σχετική οδηγία. Τώρα, δικαιοδοσία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Έχουμε το κεφάλαιο 6 του κειμένου αυτού. Εδώ ο πρώτος στόχος μας είναι να υπάρχει ομοιόμορφη εφαρμογή και ερμηνεία της Συμφωνίας Δανίας Europol. Και για να επιτευχθεί αυτό το σχέδιο κειμένου αναφέρει ότι το δικαστήριο έχει δικαιοδοσία για θέματα που αφορούν την ισχύ και την ερμηνεία της συμφωνίας αυτής που θα τεθούν από δικαστήρια της Δανίας και τα θέματα που σχετίζονται με τη συμμόρφωση της Δανίας με τη συμφωνία αυτή. Το δικαστήριο έχει επίσης αρμοδιότητα για θέματα δικαστικής προσφυγής κατά αποφάσεων ε, του επόπτη προστασίας δεδομένων και επίσης έχει αρμοδιότητα για να αποφαθεί επιθεμάτων που αφορούν η πετιότητα της Europol. Τώρα να αναφέρω και κάτι άλλο, επίσης πολύ σημαντικό, μία άλλη ρήτρα που περιέχει αυτό το σχέδιο κειμένου που αποφασίστηκε με βάση τη γνώμη του Κοινοβουλίου στην οποία προαναφέρθηκα Πρόκειται για τις διατάξεις ε, αξιολόγησης που αναφέρονται στο άρθρο 25. Τι λένε λοιπόν αυτές οι διατάξεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το αργότερο μέχρι την 31η ε, Δεκάτου 20 θα κάνει λοιπόν μία αξιολόγηση για την αποτελεσματικότητα της συμφωνίας, την λειτουργική, την επιχειρησιακή ε, αποτελεσματικότητα, καθώς και τη συμμόρφωση της Δανίας με της ρήτρα προστασίας των δεδομένων που περιέχει. Φυσικά αυτή η αξιολόγηση θα αποσταλεί και στο Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο. Και με βάση αυτή την αξιολόγηση μπορεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέχρι την 34 ε, του 2021 μπορεί να κάνει συστάσεις προς το Συμβούλιο για μια απόφαση που να επιτρέψει την έναρξη διαπραγματεύσεων που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε μια συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Δανίας που θα αντικαθιστούσε το κείμενο που συζητάμε σήμερα, την Συμφωνία Europol Δανίας. Αυτά. Γιατί θεωρώ ότι η Europol θα πει περισσότερα. Ευχαριστώ πολύ ο Πρόεδρος, ο κύριος Νιούμαν από την Europol. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καλημέρα στα αξιότιμα μέλη. Η συμφωνία αντανακλά τη συγκεκριμένη κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η Δανία μετά από την 1η Μαΐου. Αφενός ε, η Δανία είναι βεβαίως ε, κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά αφετέρου δεν ε, συμμετέχει στον κανονισμό της, Ευρωπόλ. Αυτό οδηγεί σε μια κατάσταση που είναι αντίστοιχη με άλλες τρίτες χώρες μη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διότι η Δανία θα χάσει την άμεση πρόσβαση στα συστήματα της Ευρωπόλ, θα χάσει το ρόλο της ε, και δεν θα συμμετέχει στη διακυβέρνηση της Ευρωπόλ. Δεν θα μπορεί λοιπόν να ψηφίσει στο Διοικητικό Συμβούλιο και στις διάφορες υποομάδες και θα ε, θεωρείται και μάλιστα όσον αφορά την επιχειρησιακή της συμμετοχή ως ε, μία ακόμα τρίτη χώρα ε, της οποίας η συμμετοχή στις επιχειρησιακές ε, ε πτυχές απαιτεί συγκατάθεση όλων των ε, κρατών μελών. Η κατάσταση λοιπόν στην οποία έχει περιέλθει η Δανία αναφέρεται στα εξής. Η Δανία θα πρέπει να πληρώνει συνεισφορά, η οποία είναι αντίστοιχη ίση της ε, ε, συνεισφοράς ε, που πληρώνει βάσει του ΑΕΠ της στον Ευρωπαϊκό Προϋπολογισμό. και θα πρέπει να καταβάλει και το τίμημα για να στελεχώνει τις υπηρεσίες που παρέχονται 24 ώρες το 24ωρο στην Ευρωπόλ. Επίσης θα πρέπει να εφαρμόσει και το πλαίσιο προστασίας δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα πρέπει να δεχτεί ότι η συμφωνία αυτή υπόκειται και σε έλεγχο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μετά από πέντε χρόνια από τη θέση σε ισχύ της. Αυτές οι επιπλέον προϋποθέσεις λοιπόν ε, τις οποίες ε, υποχρεούνται να τηρούν άλλα τρίτα μέρη θα καλύπτονται και από κάποια άλλα επιπλέον στοιχεία τα οποία αφορούν τη λεγόμενη Συμφωνία Νορβηγία-ΣΥΝ. Θα υπάρχουν δηλαδή και κάποια επιπλέον ωφέλη. Ε, το πρώτο είναι ότι η Δανία θα έχει μια υπηρεσία με εμπειρογνώμονες οι οποίοι θα μιλούν δανέζικα 24 ώρες το 24ωρο, είτε μέσω από της Ευρωπόλ, είτε στην Κοπενχάγη, ε, βάσει και της απόφασης που θα λάβει το Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπόλ. Δεύτερον, η Δανία θα γίνει παρατηρητής στο Διοικητικό Συμβούλιο της ε, Ευρωπόλ και στις υποομάδες, αλλά όπως σας είπα και προηγουμένως δεν θα έχει δικαίωμα ψήφου. Τρίτον, θα παραμείνει συνδεδεμένη ε, στα υφιστάμενα προγράμματα ανάλυσης στα οποία ήδη είναι συνδεδεμένη και τέλος θα ενημερώνεται άμεσα για οποιασδήποτε πληροφορίες την αφορούν. Αυτά είναι τα τέσσερα βασικά μέτρα τα οποία αποτελούν τις επιπλέον προϋποθέσεις οι οποίες καθορίστηκαν για τη Δανία στη Συμφωνία. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ και τώρα να δώσουμε το λόγο στον εισηγητή μας, τον κύριο Ντιέθ Μέρα. παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ και το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Ευρωπόλ για τις παρουσιάσεις τους. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχω και πολλά να προσθέσω, διότι είναι προφανής ε, η δέσμευση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθώς επίσης και του εισηγητή σας, να βρεθεί μια νομική λύση στην κατάσταση της Δανίας και της σχέσης της με την Ευρωπόλ. Δεν θα ήθελα να κάνω κανένα σχόλιο ε, στις παρεμβάσεις ε, που ακούσαμε προηγουμένως, αλλά θα ήθελα να καθησυχάσω σε διοργανικό επίπεδο ε, και να αναφερθώ σε κάποια συγκεκριμένα θέματα. Το θεματολόγιο δηλαδή που προτείνει ο υποφαινόμενος. 30 Μαρτίου, 5η, θα εξετάσουμε την έκθεση εδώ στην Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών. 5 Απριλίου, προθεσμία για κατάθεση τροπολογιών. 11 ή 12 Απριλίου. Με την άδειά σας κύριε Πρόεδρε, ψηφοφορία εδώ στην Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών και 27 Απριλίου, 5 5η ψηφοφορία στην Ολομέλεια. Και μια επενθύμηση. Όπως γνωρίζετε, στις 14 Φεβρουαρίου ψηφίστηκε στην Ολομέλεια η απόφαση του Συμβουλίου για να συμπεριληφθεί η Δανία στον κατάλογο των τρίτων χωρών με τις οποίες μπορεί να έχει ε, συμφωνίες συνεργασίας η Ευρωπόλ. Και το αποτέλεσμα αυτής της ψηφοφορίας είναι αδιαμφισβήτητο. 632 ψήφοι υπέρ και 10 κατά. Άρα υπάρχει σαφέστατα υποστήριξη του Κοινοβουλίου για να μπορέσει η Δανία να ε, συνεχίσει να έχει τις σχέσεις που χρειαζόμαστε με την Ευρωπόλ. Είπα τότε και επαναλαμβάνω τώρα ότι η Δανία είναι απαραίτητη για την ασφάλεια των Ευρωπαίων και για την ασφάλεια των Δανών. Τίποτα άλλο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστούμε κύριε Δίας Δεμέρα. Μόνο μία συνάδελφος ζήτησε το λόγο, η κυρία Ζίπελ. Α, έχουμε και πολλούς δανούς, δεν ξέρω αν θέλουν να μιλήσουν. Να το δηλώσουν αν το επιθυμούν. Η Μπυργκίτε Ζίπελ. Ευχαριστώ. Καταρχήν να ζητήσω συγγνώμη εκ μέρου του συναδέλφου Κατερίνα Τσινίτσι που είναι σκιώδη συγγήτρια για το θέμα αυτό και δυστυχώ κολλείεται και δεν μπόρεσα να παραστεί σε αυτή τη σημαντική ανταλλαγή απόψεων. Πάντω, ευχαριστεί τον εισηγητή Δία Δεμέρα για την προσήλωσή του σε αυτό το θέμα και αναγνωρίζουμε και τι προσπάθειε που κατέβαλε η Δανία για να εφαρμόσει το νέο κεκτημένο για την προστασία των δεδομένων. Ε, τέλη του 2015 με δημοψήφισμα η Δανία αποφάσισε από την 1η Μαΐου να εγκαταλείψει την Ευρωπόλ και παρόλο που Λυπούμαστε για την έκβαση του δημοψηφίσματος. Φυσικά οφείλουμε να σεβαστούμε ε, στο μέγιστο βαθμό την απόφαση του δανέζικου λαού. Βέβαια, δημιουργεί ένα προηγούμενο έτσι σε ό,τι αφορά την ε, συμμετοχή των κρατών μελών στου ευρωπαϊκού οργανισμού. Και όταν αποφάσισε να εγκαταλείψει την Ευρωπόλ, ε, παρόλα αυτά εξακολουθεί να είναι πλήρε μέλο Ευρωπαϊκή Ένωση. Βέβαια, όλοι συμφωνούμε ότι η επίσημη ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών ε, έχει κέρια σημασία για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος και της τρομοκρατίας και ως εκ τούτου θα πρέπει να ε, διασφαλιστεί. Παρ' όλα αυτά, εμείς ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ήδη εκφέραμε την θέση μας στο ψήφισμα σε ό,τι αφορά την ε, ένταξη της Δανίας στον κατάλογο τρίτων χωρών με τις οποίες η Ευρωπόλ μπορεί να συνάψει συμφωνίες συνεργασίας και στο ψήφισμα ζητήσαμε ρητά μία πενταετή προθεσμία προκειμένου να εξασφαλιστεί μια μεταβατική περίοδος ώστε μετά το πέρας της είτε να έχουμε μετα το περας ειτε συμμετοχή είτε μια κανονική διεθνή συμφωνία δυνάμει το άρθρο 218 της Συνθήκης Λισαβόνας, ώστε να έχουμε μια πραγματικά νομικώς ε, άρτια συνεργασία μεταξύ Ευρωπόλ και Δανίας. Και λυπούμαστε που οι συστάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δεν ελήφθησαν υπόψη από τους διαπραγματευτές της συμφωνίας αυτής. Η συμφωνία θα πρέπει να εξασφαλίζει ότι η κατάσταση αυτή έχει μόνο μεταβατικό και προσωρινό χαρακτήρα. Θα προτιμούσαμε φυσικά μια πλήρη συμμετοχή της Δανίας στην Ευρωπόλ ή την διαπραγμάτευση μιας κανονικής διεθνούς συμφωνίας που να εξασφαλίζει την ομιμότητα και των σχέσεων μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών μελών και των ευρωπαϊκών οργανισμών. Επίσης, να προσθέσω και μερικά προσωπικά σχόλια σε αυτό το θέμα. Δεν θα επαναλάβω όσα ήδη διατύπωσα στην πρώτη ανταλλαγή απόψεων που είχαμε στην Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών για το θέμα αυτό, αλλά εμένω πραγματικά σε όλα όσα είπα πέραν του του ε, είμαι βεβαία ότι όλοι μας ε, έχουμε την προθυμία να πραγματοποιήσουμε τα απαραίτητα βήματα και τις ενέργειες ώστε να συνεχίσουμε την ίδια αγαστή συνεργασία που υπάρχει μεταξύ Δανία και Ευρωπόλ. Παρόλα αυτά, ε, με μπερδεύει κάπως και με θλίβει αυτή η κατάσταση, γιατί νομίζω ότι δεν έχουμε την ε, τη δέσμευση όλων των συμμετεχόντων για μία, αν μη τι άλλο, σαφή και άρτια διεθνή συμφωνία. Δεν βλέπουμε στο προτινόμενο σχέδιο συμφωνίας ένα ξεκάθαρο χρονοδιάγραμμα που θα οδηγήσει σε μια κανονική διεθνή συμφωνία, που είναι η ελάχιστη προϋπόθεση για μας. Και ταυτόχρονα θέλουμε μεγαλύτερη συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και επίσης ε, σαφέστερες διακηρύξεις και δεσμεύσεις των ε, ενδιαφερομένων, ώστε να βοηθήσουμε τη Δανία να βρει μια κατάλληλη λύση και ε, να ξαναγίνει η Δανία σε τελική ανάλυση πλήρες μέλος της Ευρωπόλ. Ευχαριστώ. Κύριος Βίστερσεν. Εγώ θα μιλήσω δανέζικα. Σας ευχαριστώ. Η συμφωνία για την ε, σύνδεση τη Δανία με την Ευρωπόλ στο μέλλον είναι πολύ σημαντική, όχι μόνο για την Ευρωπόλ, αλλά και για την ίδια τη Δανία. Και μείναμε πολύ ικανοποιημένοι από την πορεία της διαδικασίας. Και έτσι η Δανία θα υποφεληθεί από πολλά επιχειρησιακά ωφέλη με τη συνέχιση αυτής της συνεργασίας και θα συμβάλλει στην καταπολέμηση σοβαρού εγκλήματος και τρομοκρατίας στην Ευρώπη. Η ομάδα μεταρρυθμιστών και συντηρητικών και το Δανέζικο Κόμμα των Λαών που εκπροσωπώ ε, είναι υπέρ αυτής της ενισχυμένης συνεργασίας με όσο το δυνατό λιγότερα προσκόμματα και ενδιασμούς για τη μελλοντική συνεργασία. Ελπίζω να μην ε, υποστούμε περιτές πιέσεις, γιατί υπάρχει σαφή δέσμευση όλων των ενδιαφερομένων Συμβουλίου ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Δανίας να παραμείνει η Δανία ε, ενεργός παράγων της ευρωπαϊκής ασφάλειας. Αυτό γινόταν μέχρι τώρα και θέλουμε να συνεχιστεί. Και είμαστε κατά ρητρών, όπως της ρήτρας σταδιακής εκπνοής ή του εσωτερικού μηχανισμού αξιολόγηση. Ο κύριος Πίτερσον και εγώ θα μιλήσω δανέζικα επίση. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω θερμά τους συναδέλφους της Επιτροπής και φυσικά και τον εισηγητή μας, τον κύριο Αγκουστίν Διασδεμέρα, που απέδειξε ότι μπορούμε να κατηγορούμε μερικές φορές τις Βρυξέλλες ε, ε, για γραφειοκρατία και χρονοβόρες διαδικασίες, αλλά αυτή τη φορά χάρη στην ε, σπουδή των συναδέλφων και στην προθυμία τους ε, διεκπεραιώνουμε σχετικά γρήγορα αυτό το ζήτημα. Φυσικά δεν είναι προς το κοινοτικό συμφέρον ε, η Δανία ε, και τη μικρή χώρα να δημιουργήσει πρόβλημα ή κενό ασφάλεια στην υπόλοιπη Ευρώπη. Η Ευρωπόλ είναι σήμερα το κέντρο το συντονιστικό κέντρο της συνεργασίας που έχει κέρια σημασία στην υπολοιπη ευρωπη η Ευρωπόλη ειναι σημερα το κεντρο το συντονιστικο κεντρο της συνεργασιας που εχει κερια σημασια στην καταπολεμηση του οργανωμένου εγκλήματος. Πριν από ένα μόλις χρόνο είχαμε την τρομοκρατική επίθεση στην Ευρώπη και η τρομοκρατική απειλή συνεχίζεται στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο και στις ευρωπαϊκές πόλεις. Δεν μπορούμε λοιπόν να έχουμε αδύναμους κρίκους στη συνεργασία μας, ούτε στην προστασία των εξωτερικών μας συνόρων, ούτε στην προστασία και ασφάλεια των πολιτών μας. Και η συμφωνία αυτή δίνει στη Δανία μία πρόσβαση στη βάση δεδομένων που δεν είναι πλήρης, αλλά είναι επαρκής. Και εγώ θα προτιμούσα να είμαστε πλήρες μέλος η Δανία της Ευρωπόλ, δεν το κρύβω, αλλά μια και δεν μπορούμε να παραμείνουμε πλήρη μέλη, δεν μπορούμε να έχουμε και την ίδια πρόσβαση και τα ίδια ωφέλη από τη συνεργασία ε, με την Ευρωπόλ όπως οι υπόλοιπε χώρες που είναι πλήρη μέλη. Γι' αυτό και πιστεύω ότι θα πρέπει να είναι χρονικά περιορισμένη αυτή η συμφωνία μεταβατική και να γίνει σύντομα αναθεώρησή της όπως προβλέπει και το κείμενο. Επίσης, να δούμε και το θέμα της αξιολόγησης από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Χαίρομαι που θα κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την αξιολόγηση, αλλά όχι ερήμην του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θα πρέπει και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να λάβει ενεργό μέρο σε αυτή την αξιολόγηση, ώστε με ανοιχτό, δημοκρατικό και διαφανή τρόπο να πραγματοποιηθεί η αξιολόγηση τη συμφωνία. Και σα ευχαριστώ για την ευχάριστη αυτή συνεργασία που είχαμε. Ωραία, ευχαριστώ κύριε Ντεμέρα, Αν δεν θέλει κανείς άλλος να πει κάτι, δεν ξέρω αν θέλετε κύριε Διαθδεμέρα να αντιδράσετε σε αυτά που αναφέρθηκαν και εγώ θα ήθελα, αλλά όχι λέει ο κύριος Διαθδεμέρα, δεν θα απαντήσω. Να ευχαριστήσω για την επικοδομητική στάση των συναδέλφων για να, να υπερβούμε αυτήν την ε, νομικά πρωτότυπη κατάσταση. Δεν θέλει κανείς άλλο το λόγο. Ωραία. Πριν αναφερθώ στα πρακτικά θέματα, τα οποία ανέφερε και ο κύριος Δίας Δεμέρα, να αντιδράσω και εγώ σε αυτά που είπε η Μπίργκη Τζίπελ, το ευρύτερο ζήτημα που θα πρέπει να τονίσουμε πριν δούμε το σχέδιο έκθεση είναι ότι υπάρχουν αρμοδιότητες του Κοινοβουλίου για το θέμα αυτό. Ο κύριος Ντεμέρα είναι μετριοπαθής και μετριόφρον. Αλλά πρέπει να έχουμε υπόψη τις αρμοδιότητές μας. Η συμφωνία αυτή από την ίδια της τη φύση δεν μπορεί να είναι τέλεια, το καταλαβαίνουμε. αλλά υπάρχει ευρεία πολιτική συνένεση ότι η Δανία θα πρέπει να συμμετέχει στην ε, Ευρωπόλ. Πρέπει λοιπόν να κάνουμε ό,τι μπορούμε, ούτως ώστε να έχει την καλύτερη δυνατή παρέμβαση το Κοινοβούλιο. Θα έχουμε την έκθεση, συγγνώμη, πρώτα την ε, αξιολόγηση και μετά θα έχουμε και μια έκθεση από την ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ κύριε Ντίαθ Μέρα που είστε ιδιαίτερα προσεκτικός. Αλλά καταλαβαίνω και τις ανησυχίες που έθιξε η κυρία Ζίπελ και υπάρχει ευρεία πολιτική στήριξη για να συμμετάσχει η Δανία στην Ευρωπόλ εκφράστηκε σαφώς και σήμερα. Λοιπόν, τώρα το σχέδιο έκθεση θα υποβληθεί στις 30 ε, Μαρτίου, αρχές Απριλίου θα έχουμε την ε, προθεσμία υποβολής τροπολογιών, μάλλον 5 Απριλίου η ψηφοφορία θα μπορούσε να γίνει στις 11 ή 12 Απριλίου όπως υπενθύμησε ο κύριος Δίας και στοχεύουμε να ψηφιστεί στην Ολομέλεια τον Απρίλιο. Εντάξει. Ευχαριστώ πολύ. Οπότε κλείσαμε αυτό το θέμα. Να περάσουμε στο 16 που είναι οι συνθήκες ε, υποδοχής στα πλαίσια του κοινού ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου. Μετά την παρουσίαση του σχεδίου έκθεση από την Σοφία Ιντφελ τον Ιανουάριο, όταν είχαμε μια συζήτηση για θέματα όπως η πρόσβαση στην αγορά εργασίας, ε, μαθήματα γλωσσών, τύποι προσέγγισης ε, για τις δευτερογενείς μετακινήσεις και την μεταχείριση των ευαλώτων προσώπων, ιδιαίτερα των ανηλίκων. Τώρα μπορούμε να κάνουμε μια ανταλλαγή απόψεων για τις 491 τροπολογίε που υπευλήθησαν. Τώρα θα δώσω το λόγο στην εισηγήτριά μας για να σχολιάσει τις τροπολογίες και να μας ενημερώσει για το θέμα αυτό. Σοφή, έχεις το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Κλοντ. Θα είμαι πολύ σύντομη. Είχαμε περίπου 500 τροπολογίες. Αυτή τη στιγμή εκπονούμε συμβιβαστικέ. Είχαμε δύο μακροσκελείς συνεδριάσεις των συντονιστών και ήδη συμφωνήσαμε επί αρκετών συμβιβασμών. Έχουμε ακόμη ορισμένους ε, υπό αλλά είμαι σχεδόν σίγουροι ότι θα καταλήξουμε σε συμβαστικές τροπολογίες για τα περισσότερα θέματα που θα στηριχθούν, ας πούμε, από την πλειονότητα των πολιτικών ομάδων, όχι από όλες. Κάποιες τροπολογίες που υποβλήθηκαν, παρά το ότι τις σέβομαι, είναι εντελώ αντίθετες από το πνεύμα της έκθεσης, άρα δεν μπορούν να συμπεριληφθούν σε συμβασμούς, αλλά έτσι λειτουργεί η δημοκρατία, θα πρέπει ακριβώς να τις ψηφίσουμε. Θα υπάρξουν λοιπόν συμβιβασμοί για τους ορισμούς, για το πεδίο εφαρμογής, την ε, πληροφόρηση που πρέπει να δίνεται στους ετούμενους. Μισό λεπτό, Σοφή. Συνάδελφοι, σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ, συνεχίστε τη συνεδρίαση. Ευχαριστώ πολύ. Μήπω μπορείτε τις συζητήσεις να τις κάνετε έξω, παρακαλώ Σοφή. Για θέματα λοιπόν, λέει η κυρία Ινφέλντ, κράτηση, όπως κράτηση, το δικαίωμα ε, μετάβαση σε άλλα κράτη-μέλη ή και τρίτες χώρες, πρόσβαση στην αγορά εργασία, ε, μαθήματα γλωσσών, ε, κατάρτιση για τα πολιτικά δικαιώματα, κατάσταση των παιδιών, ειδικέ ανάγκες υποδοχής, η ε, υγειονομική κάλυψη, όλα αυτά τα θέματα τα συζητάμε. Σε ορισμένα ακόμη δεν έχουμε συμφωνήσει, αλλά στα περισσότερα έχουμε. Δεν μπορούμε φυσικά να αποφασίσουμε 100% για κάθε λεπτομέρεια, γιατί πρέπει να λάβουμε υπόψη και διάφορους άλλους κανονισμούς και τους κανόνες του Δουβλίνου είναι κάπως περίπλοκο, αλλά προχωράει. Και όπως σας είπα, είμαι ε, σίγουρη, είμαι αρκετά σίγουρη θα έλεγα, ότι μπορούμε να επιτύχουμε συμφωνία για τα περισσότερα θέματα. Ωραία. Οι συντονιστές. Ο κύριος Πουλιέζε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχάς ε, θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για την προσπάθειά της και την απόπειρα να προσπαθήσει να συγκεράσει τις διάφορες πολιτικές απόψεις, κάτι το οποίο δεν είναι εύκολο, όπως είπε και η ίδια στην εισαγωγή της. Εμείς συμφωνούμε με κάποιες από τις επιλογές που έγιναν κυρίως ε, το γεγονός ότι πρέπει να υπάρχει μία δικαστική αρχή και να μην υπάρχει διοικητική αρχή αρμόδια για τα στοιχεία τα οποία περιορίζουν την ε, ατομική ελευθερία, για τα δικαιώματα των ανηλίκων, ε, τα μαθήματα γλωσσών, την διαδικασία αγωγής του πολίτη για να βοηθήσουμε την ένταξη αλλά ε, υπάρχουν και κάποια θέματα για την πρόσβαση στην αγορά εργασίας, ε, ε, κυρίως όσον αφορά στην άμεση πρόσβαση, με την οποία διαφωνούμε. Όσον αφορά την διαπραγματευτική τακτική, την οποία συζητήσαμε σε μια συνεδρίαση των σκιωδιών εισηγητών, δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε με την επιλογή και θα θέλαμε επίσης να διαφυλάξουμε και κάποια πράγματα τα οποία είπαμε στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Άρθρο 15, παράγραφος 2, 2 εκεί προτείνεται διαγραφή όπου λέγεται ότι για λόγους που σχετίζονται με τα όρια της αγοράς εργασίας τα κράτη-μέλη πρέπει να επιβεβαιώσουν κατά πόσον μία ε, θέση θα πρέπει να πληρωθεί πρώτα από κράτος μέλος της, ε, από ε, υπήκο της χώρας. Και επίσης έχουμε την τροπολογία 357 όπου λέγεται ότι οι εθνικές αρμόδιες αρχές σε συμφωνία με τις τοπικές αρχές μπορεί να ευνοούσουν την απασχόληση ατόμων που χρήζουν ε, ε, προστασίας διεθνούς ε, βάσει των ανθρώπων που βρίσκονται εκεί θεωρούμε ότι αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια διαδικασία καλύτερης ένταξης. Υπάρχει μια πρόταση ε, συμβιβαστική η οποία έχει επισημοποιηθεί αλλά ε, δεν μας ικανοποιεί διότι είναι πιο ήπιο από αυτό το οποίο θα θέλαμε. Ευχαριστώ η Κέιτη Πύρη από τους Σοσιαλιστές και Δημοκράτες. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Γελάνε για το όνομά μου εδώ. Θα ήθελα να υποστηρίξω την εισηγήτρια, διότι θέλει να επικεντρωθεί σε θετικά κίνητρα και όχι σε μέτρα τιμωρίας ε, για να βοηθήσει και να βελτιώσει και την ε, ε, υποδοχή στα κράτη-μέλη. Αυτό σημαίνει ότι θα έχουν τη δυνατότητα οι αιτούντες άσυλο να μεταφερθούν σε άλλη χώρα. Επίσης ε, βλέπουμε ότι υπάρχει μεγάλη πολιτική υποστήριξη να διαγραφεί η δυνατότητα να κρατούνται παιδιά από τα κράτη-μέλη απλώς και μόνο γιατί κάνουν αίτηση ασύλου. Μια άλλη βελτίωση στην πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι σαφεί ορισμοί, καλύτερε δικλείδε ασφαλεία για τα θεμελιώδη δικαιώματα, βελτίωση στη νομική συνδρομή και ε, μαθήματα βοήθεια ένταξη, όπω για παράδειγμα μαθήματα γλωσσών από την πρώτη μέρα. Η μόνη επιφύλαξη που θα ήθελα να θίξω είναι η προσωρινή πρόσβαση στην αγορά εργασία. Παρά το γεγονό ότι αντιλαμβάνομαι ότι το να μπορεί κάποιο να δουλέψει είναι ο καλύτερο τρόπο να ενταχθεί στην κοινωνία, θα πρέπει ε, να μην επιτρέψουμε κατάχρηση του συστήματος ασύλου και να μην χρησιμοποιείται ως ε, πρόσβαση για τους οικονομικούς μετανάστες θα πρέπει να παρέχεται ε, δυνατότητα εργασίας όντως το αργότερο 9 μήνες μετά την ένταξη. Ε, εμείς προτείνουμε μείωση στους 6 μήνες και η συγκήτρια και κάποιοι άλλοι προτείνουν πρόσβαση στην αργά εργασίας από την πρώτη ημέρα ε, που γίνεται η αίτηση ασύλου. Επειδή όμως υπάρχουν πολλοί αιτούντες που δεν θεμελιώνουν την ε, δυνατότητα χορήγησης ασύλου. Έρχονται, θέλουν να εργαστούν κάποιες ε, μήνες και μετά επιστρέφονται στη χώρα καταγωγής τους. Ε, και αυτό σημαίνει ότι υπάρχει δυνατότητα να εργάζονται για τους λάθους λόγους. Υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι βρίσκονται στην ταχεία διαδικασία και όντως δεν έχουν πρόσβαση στην εργοσίες αλλά μπορεί να προκύψει να ισχύει η διαδικασία για κάποιον αργότερα από τη ε, τη στιγμή που κατέθεσε την ε, αίτηση. Εμείς λοιπόν προτείνουμε η πρόσβαση στην αγορά εργασίας να δίνεται μετά την ε, ταχεία διαδικασία και όταν οριστικοποιηθεί, δηλαδή μέσα σε ένα διάστημα δύο μηνών. Αυτό μας εγγυάται ότι μόνο αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι κατά πάσα πιθανότητα θα λάβουν το άσυλο θα μπορέσουν να ενταχθούν στην αγορά εργασία και αυτό αποτελεί ε, και πάρα πολύ κίνητρο, ε, καλό κίνητρο για ταχύτερη ένταξη. Προσβλέπω στη συνεργασία για το θέμα αυτό με την εισηγήτρια και του Σκιώδη. Το κύριο Αλαχάχο από το ECR. Ευχαριστώ. Θα ήθελα καταρχήν και εγώ να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για την πολύ φιλόδοξη στάση της και την αργότερη προσπαθειά της. Δυστυχώς η δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε με την προσέγγιση της και τις προτινόμενες συμβαστικές τροπολογίες. Γιατί έχουμε εκτεταμένη χρήση του συστήματος ασύλου ως ε, πρόσχημα από τους οικονομικούς μετανάστες αφενός και έχουμε και δευτερογενείς μετακινήσεις και αναζήτηση της ευνοικότερης χώρας για χορήγηση ασύλου από την άλλη. Δεν Θέλουμε να αποθαρρύνουμε τους, τους μετανάστες ε, να παίρνουν τη Μεσόγειο και να έχουμε κάποια ανάπτυξη ότι αυτού που πραγματικά είναι νομοταγεί και τηρούν του κανόνε. Θα πρέπει να έχουν ε, δικαίωμα οι αιτώντε άσυλο, όχι το δικαίωμα να μην συνεργάζονται, να ψεύδονται ή να παραβιάζουν ατιμόρυτα του κανόνε. Θα πρέπει να βρούμε την ισορροπία μεταξύ των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων. Θα πρέπει να εναρμονίσουμε τα πρότυπα και τι προδιαγραφέ μα, αλλά εναρμονισμένα πρότυπα θα πρέπει να είναι ρεαλιστικά για όλα τα κράτη-μέλη. Και από οικονομική άποψη, αλλά και από άλλες απόψεις. Και όταν είναι υπερβολικά γενναιόδωρα και φιλόδοξα τα πρότυπα, ε, δεν θα τηρηθούν και κάποιες χώρες θα είναι πιο ελκυστικές ε, για τους μετανάστες από άλλες. Και παρόλο που είμαστε υπέρ της πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ε, έχουμε κάποια θέματα ακόμη και σίγουρα το σχέδιο έκθεσης δεν μας ικανοποιεί. Ε, επίσης υπάρχει δυνατότητα κράτησης των ετούντων, για να αποφευθεί η δραπέτευσή του η εξαφάνισή τους. Βέβαια, η συμβαστική τροπολογία παρα... περιορίζει αυτή τη δυνατότητα και στην πράξη είναι αδύνατο για τις αρμόδιες αρχές να αποδείξουν ότι ένας ετών θα εξαφανιστεί. Μόνο κατόπιν ορτής γίνεται η διαπίστωση απλώς της εξαφάνισής του. Και πολύ προβληματική είναι η κατηγορηματική απαγόρευση της κράτησης ε, ανηλίκων. Ε, βέβαια, αυτό ισχύει και για παιδιά που είναι σχεδόν στο όριο τη ενηλικίωση ή κάποιου που ισχυρίζονται την ανήλικη χωρίς χωρί να είναι. Και μάλιστα από άποψη δημόσια τάξη, αυτή είναι και πιο περίπλοκη ομάδα ε, και επικίνδυνη και είναι ένα από του ε, εύλογου λόγου για την κράτηση. Επίση, ε, στα κράτη-μέλη σχεδόν όλοι οι ανήλικοι ε, για τους οποίους έχουν απορριφθεί αίτηση άσυλο εξαφανίζονται. Επίσης, δεν μας αρέσει να ε, ε, επεκτείνουμε διαρκώς τον κατάλογο με τους ετούντες ειδικής προστασίας, ειδικών αναγκών. Ε, μιλούμε για τους αναπήρους, ε, τα παιδιά και θεωρούμε ή τα, τους, τα θύματα βασαριστήριων να συμπεριλαμβάνονται, αλλά αναφέρονται και οι τα έφηβα κορίτσια, οι, οι ελεύθερες γυναίκες, ΛΟΑΔΜ, άπιστοι, με θρησκευτικές μειονότητες. Νομίζω ότι είναι υπερβολικά διαβριμένος αυτός ο κατάλογος με τους μετανασμίδικες ανάγκες. Επίσης, η βασική Τροπολογία 19 απαγορεύει κατηγορηματικά την κράτηση ετούντο που έχει ειδικέ ανάγκες υποδοχής. Οπότε ουσιαστικά γίνεται αδύνατη κράτηση οποιοδήποτε, ακόμη και όταν ε, οι συνθήκες απαιτούν μια τέτοια κράτηση. Θέλουμε επαρκείς κυρώσεις για τους ετούντες που εξαφανίζονται από, το, από τον τόπο ε, παραμονής τους ή δεν πληρούν ε, τις, ε, την υποχρέωση της παρουσίασής τους ή παραβιάζουν τους κανόνες. Το άρθρο 19, παράγραφος 1, προβλέπει μείωση ή αναστολή της ε, ημερήσιας αποζημίωσης σε, τέτοια προϋπόθεση, σε τέτοιες περιπτώσεις. Η Συμβαστική Τροπολογία 17 όμως λέει ότι ενώ με εξασφαλίζει, ε, θα πρέπει ε, να εξασφαλίζει ένα κατάλληλο βιωτικό επίπεδο. Νομίζω ότι με μια τέτοια συμβαστική τροπολογία καταργούμε το αποτρεπτικό χαρακτήρα της κύρωσης. Εγώ, ως πολίτης χώρας μου, μπορώ να χάσω τα κοινωνικά επιδόματα που δικαιούμαι αν δεν πληρώ κάποιες στοιχειώδεις ε, υποχρεώσεις μου. Θα πρέπει το ίδιο να ισχύει και για τους ετούντες άσυλο. Γιατί δεν είναι παράλογες οι απαιτήσει αυτές, ούτε υπάρχει εύλογος αποχρολόγος ε, να τους παραβιάζει ένας ετών άσυλο. Αυτά κύριε Πρόεδρε. Έχουμε καταθέσει αρκετές τροπολογίες με στόχο να δώσουμε έμφαση το καθήκον των ετούντων να διευκολύνουν τις αρμόδιες αρχές και το γραφειοκρατικό άκθος τους και να καταστήσουμε το σύστημα ασύλου λιγότερο ελκυστικό για αυτούς που δεν χρήζουν πραγματικά προστασίας. Ελπίζω να εξετάσει τις τροπολογίες μας η κυρία εισηγήτρια και ενδεχομένω να τις υποστηρίξει κιόλα. Ευχαριστώ. Καταρχάς, στον προηγούμενο μιλτή να πω ότι πρόκειται με οδηγία υποδοχής, όχι μια οδηγία αποτροπής. Είναι κάποια μικρή διαφορά στον τρόπο αντιμετώπισης. Φυσικά η Ευρωπαϊκή Ένωση συνειδητά αποφασίστηκε πριν έρθουμε εμείς εδώ να υπάρχει μια οδηγία υποδοχής, υποδοχής προσφύγων, για να ρυθμίσουμε τα θέματα αυτά τώρα συζητάμε, όχι κάτι άλλο. Δεν χρειάζεται να συζητάμε λοιπόν το στόχο. Νομίζω λοιπόν ότι αυτό το οποίο έχουμε ενώπιόν μας αν μας επιτρέψει να βελτιώσουμε έστω και λίγο τις συνθήκες ζωής των προσφύγων που έρχονται σε μας, θα είχε θετικό αποτέλεσμα. Και νομίζω ότι είναι θετικό το ότι η συγγήτρια έλαβε υπόψη πολλά από αυτά τα οποία λένε ε, πολλές μη και ο μικρόν, αλλά και διάφορα κράτη-μέλη. Τώρα για τα διάφορα σημεία αυτές οι ειδικέ ομάδες που έχουν αναφερθεί ε, πολλές φορές είναι καλό να πούμε ότι είναι άτομα που έχουν ειδικέ ανάγκες. Αυτές είναι οι ομάδες. Αυτό πρέπει να κοιτάξουμε. Γιατί πρέπει να κάνουμε συγκεκριμένες διαφοροποίησεις. Είναι ορισμένες ε, ε, άγαμες γυναίκες που δεν έχουν δεν δικαιούνται αυτές τις ειδικέ ανάγκες. Αλλά υπάρχουν διάφορες ε, άγαμες γυναίκες οι οποίες υπέστησαν τρομερά κατά τη, δεινά κατά τη διάρκεια της πορείας τους. Για παράδειγμα από το Ιράκ έχουμε πολλές γυναίκες οι οποίες εκεί υπέστησαν ε, τέτοια δεινά από τον ΤΑΕΣ που τώρα έχουν ειδικέ ανάγκες. Επαναλαμβάνω λοιπόν, δεν σημαίνει ότι αφορούν όλα τα άτομα. Το θέμα είναι να δούμε ε, μεμονωμένα τα άτομα τι ανάγκες έχουν. Και αυτό είναι μεγάλη πρόοδος. Μέχρι στιγμής δεν έχει συμβεί. Και είναι μία από τις κυριότερες επικρίσεις ε, που έχουν διατυπωθεί τα τελευταία χρόνια. Τώρα όσον αφορά τι σημαίνει η επανένωση των οικογενειών, είναι θετικό. Θα βοηθήσει να υπάρξει και η κοινωνική ένταξη πολύ περισσότερο, σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό από ό,τι προηγουμένω. Και αυτό το θεωρώ σωστό γλωσσικά μαθήματα. Βεβαίως, βεβαίως, είναι πολύ σημαντικό να μπει στο κείμενο. Αλλά το θέμα είναι, όπως και πριν, ποιος θα πληρώσει και για τα μαθήματα γλωσσών και για άλλα. Εγώ νομίζω ε, ότι τουλάχιστον ε, τα μαθήματα γλωσσών πρέπει να είναι δωρεάν θα πρέπει ότι άλλο και αν ε, πρέπει να πληρωθεί, τα μαθήματα γλωσσών πρέπει να είναι δωρεάν. Επ' αυτού πραγματικά πιστεύω ότι πρέπει να είναι δωρεάν. Και τώρα, με τις παραγράφους 4 και 5 του άρθρου 16 έχουμε ένα πρόβλημα. Δεν νομίζουμε ότι έχουν έννοια. Γιατί εγώ δεν έχω εμπιστοσύνη ότι τα κράτη-μέλη δεν θα εκμεταλλευτούν αυτές τις ε, ρήτρε. Μπορεί να αξιοποιηθούν λοιπόν και τελικά να, καθιστούν, να καταστούν υποχρέωση. Δεν μας ικανοποιεί. Η κράτηση βεβαίως. Εμείς ως αριστερά ε, έχουμε μεγάλες διαφωνίες με την κράτηση. Βεβαίως αναφέρονται προϋποθέσεις για τους ανήλικους ότι θα πρέπει να ελέγξουμε αν υπάρχουν ειδικέ ανάγκες εκ των προτέρων. Αυτά μπορούν να θεωρηθούν ε, πρόοδος. Τώρα για την ένταξη στην αγορά εργασίας. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει καθόλου. Αν έρθει κάποιος, ε, για παράδειγμα στην δική μου περιοχή, ήρθε ένας γιατρός από τη Συρία, στη δική μου περιοχή της ε, Γερμανίας, με πολύ καλά προσόντα. Δεν μπορούσε να εργαστεί. Πρώτα απ' όλα πρέπει να μάθει γλώσσα, Πρώτα απ' όλα πρέπει να ικανοποιήσει μια σειρά υποχρεώσει. Ούτω ή άλλω όλα αυτά παίρνουν κάποιου μήνε. Και μετά βρέθηκε ένα νοσοκομείο που είπε βεβαίω τον θέλουμε, τον θέλουμε. Να κάνει μια εκπαίδευση σε εμά και μετά να τον βοηθήσουμε. Να ένα παράδειγμα είναι υψηλού επίπεδου, υψηλών προσόντων. Αλλά το βασικό είναι λοιπόν να βοηθήσουμε τους πάντες να ενταχθούν άνετα στην αγορά εργασίας. Εάν ε, χρειάζεται να περάσουν μήνες, τότε δημιουργούνται άλλες ανάγκες και πιέσεις. Δεν μπορούν να ενταχθούν. Γιατί πρέπει να μάθουν και τη γλώσσα για να ενταχθούν. Και τι άλλο, τι άλλο. Υπάρχουν και άλλα βέβαια, αλλά ίσως τα ξέχασα. Λοιπόν, καλό είναι να δούμε τι θα προκύψει σε σχέση με τον Δουβλίνο, να μην τα επιλέξουμε τώρα όλα. Με συγχωρείτε, χτυπάει και το τηλέφωνό μου. Ευχαριστώ πολύ, λοιπόν. Ε, εντάξει, θέλετε να συνεχίσετε. Νομίζω ότι καταλάβαμε πού το πάτε γενικώς και την ε, σαφή αντίθεσή σας με τον προηγούμενο μιλητή. Απλώς αναφέρομαι σε γεγονότα, δεν επιδιώκω να, να κάνω πολιτική εκμετάλλευση. Τελείωσες Κορνέλια. Νομίζω ότι καταλάβαμε τη γενική κατεύθυνση των τροπολογιών που θα υποβάλεις. Ωραία. Η Μπόντιλ τώρα, από τους πράσινους. Ευχαριστώ πολύ. Περιμένω να βάλετε και τα ακουστικά σας. Και ευχαριστώ την Σοφή για την πολύ καλή εργασία για τους συμβασμούς, για το θετικό κλίμα, το κλίμα συνεργασίας ε, μεταξύ των σκιωδών. Είναι ένα εξαιρετικά σημαντικό νομοθέτημα είναι τμήμα του πολύ σημαντικού και εκτεταμένου πακέτου για το άσυλο, το οποίο εξετάζουμε σιγά σιγά, αναθεωρώντας ε, διάφορα νομοθετήματα. Πολύ σημαντική λοιπόν οδηγία. Οι συνθήκες από χώρα σε χώρα, ξέρετε, διαφέρουν. Γι' αυτό όλοι φοβόμαστε ότι οι ετούντες θα επιλέγουν ε, τη χώρα που θεωρούν ότι είναι πιο ευνοϊκή. Δεν λέμε ότι θα γίνουν ποτέ ταυτόσιμες οι συνθήκες, αλλά θέλουμε τουλάχιστον σε κάθε κράτος μέλος να υπάρχουν κάποιες ελάχιστες προϋποθέσεις και τα κράτη-μέλη να εφαρμόσουν τα νομοθετήματα τα οποία έχουν εγκρίνει. Τώρα σε σχέση με την προηγούμενη νομοθεσία υπάρχει κάποια πρόοδος αλλά εξακολουθώ να θεωρώ ότι είναι ανεπαρκής η προβλέψεις για τα παιδιά. Δεν συμφωνούμε με αυτό. Αλλά θέλω να αναφερθώ σε κάτι που πραγματικά θεωρώ πολύ σημαντικό. Είναι οι ετούντες οι οποίοι ήδη είχαν κάποια απασχόληση αλλά χρειάστηκε να την διακόψουν. Και χρειάζεται λοιπόν να ε, ζητήσουν άδεια εργασίας και όχι άσυλο. Ορισμένοι φοβούνται ότι μπορεί να παρέχουμε υπερβολικά δικαιώματα τους ετούντες άσυλο. Στην Σουηδία το σύστημά μας είναι ως εξής. Εάν ο, ο ετών και οι αρχές θεωρούν ότι δεν είναι δυνατόν να ολοκληρωθεί η εξέταση της αίτησή του σε λιγότερο από τέσσερις μήνες, τότε τους δίδεται μία εξαίρεση και μπορούν να αρχίσουν να δουλεύουν από την πρώτη μέρα που είναι εκεί. Εάν και οι δύο πλευρές θεωρούν λοιπόν ότι θα καθυστερήσει άνω των τεσσάρων μηνών η εξέταση του αιτήματό του, της αίτησης ασύλου. Εάν ένα άτομο λοιπόν έχει εργαστεί για μια σειρά μηνών, μετά ότι μπορεί να μην ζητήσουν πλέον άσυλο, απλώς να ζητήσουν άδεια εργασίας. Και εμείς δεν διαπιστώσαμε αύξηση του αριθμού ατόμων που έρχονται στη χώρα μας λόγω αυτής της ε, δυνατότητας, αντίθετα μείωση. Μείωση των ε, ατόμων ε, που ετούνται άσυλο. Προτείνουμε λοιπόν κάτι που ίσως κάποια κράτη-μέλη να μπορούν το καθένα να επιλέγουν διαφορετικούς τρόπους αντιμετώπισης των θεμάτων αυτών, ανάλογα με τις δυνατότητές τους. Ορισμένοι είπαν δύο μήνες. Βεβαίω υπάρχουν αδικαιολόγητε ε, αιτήσει ασύλου, οι οποίε ε, θα πρέπει να απορριφθούν. Μόνο οι αιτιολογημένε θα προωθηθούν και θα εγκριθούν. Είναι σημαντικό λοιπόν αυτό. Νομίζω ότι έτσι μειώνουμε τα δεινά και τι ε, δυσκολίε. Ξέρετε, είναι δύσκολο να πάρει κανεί άσυλο. Αν είσαι από το Αφγανιστάν, δεν θα σου παρασχεθεί άσυλο. Ε, ορισμένοι μπορεί βέβαια, αλλά όχι όλοι. Και εγώ του καταλαβαίνω τους Αφγανούς που έρχονται και που ετούνται άσυλο. Γιατί έρχονται από περιοχή όπου υπάρχουν, υπάρχει σύραξη. Αλλά εμείς στην Ευρώπη τους αντιμετωπίζουμε ως οικονομικούς ε, μετανάστες. Είναι λοιπόν πολύ σημαντική αυτή η μεταρρύθμιση. Μπορούμε να ενθαρρύνουμε τα κράτη-μέλη να εισαγάγουν τέτοιου τύπου κανόνες, όπως αυτός που προανέφερα στο σύστημά μου. Υποθέτω ότι θα το συζητήσουμε και περαιτέρω το θέμα αυτό στην επόμενη συνεδρίαση των σκιωδών και είμαι σίγουρη ότι θα βρούμε μια καλή λύση. Ευχαριστώ πολύ. Ωραία, σε ευχαριστούμε πολύ. Να δώσω και πάλι το λόγο στη Σόφη τώρα για να ολοκληρώσουμε για το σημείο αυτό. Μήπως θέλετε να ακούσετε πρώτα τι έχει να πει η Προεδρία. Συγγνώμη, δεν σας ε, είδα η κυρία Μπέλα. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη, θα ήθελα καταρχάς να συγχαρώ την εισηγήτρια και τους κοιόδη εισηγητές ε, για την πολύ σημαντική πρόοδο που έχει επιτευχθεί στο θέμα αυτό και θα ήθελα και επί τη ευκαιρία να σας δώσω και κάποιες πληροφορίες ε, για την πρόοδο που έχουμε καταγράψει στις ε, ομάδες του Συμβουλίου που προετοιμάζουν το θέμα αυτό. Η πρώτη εξέταση ολοκληρώθηκε στην ομάδα εργασία ασύλου στη διάρκεια της Σλοβακική Προεδρίας και στη διάρκεια της Μαλτέζική Προεδρία εξετάστηκαν αρκετά άρθρα της οδηγίας ε, στα πλαίσια μιας θεματικής προσέγγισης ε, μαζί με τις υπόλοιπες προτάσεις για το ε, πακέτο για το άσυλο και αυτά έγιναν στα πλαίσια τριών θεμάτων εγγύησεις ε, για όσους έχουν ειδικέ ανάγκες, ε, περιορισμός των δευτερογενών μετακινήσεων και κοινωνικά και οικονομικά δικαιώματα ετούντων άσυλο και ε, άτομων που δικαιούνται διεθνούς προστασίας. Ένα αναθεωρημένο κείμενο συζητήθηκε στην Ομάδα Εργασίας Ασύλου στις 16 Μαρτίου και στη διάρκεια αυτής της συζήτησης προέκυψε ότι υπάρχει σύγκληση πλέον σε αρκετές πτυχές της πρότασης, Ωστόσο, υπάρχουν κάποια σημαντικά στοιχεία τα οποία πρέπει να συζητηθούν περαιτέρω, κυρίως ε, θέματα που αφορούν την πρόσβαση των ετούντων άσυλο στην αγορά εργασίας και μέτρα για την πρόληψη των δευτερογενών ε, μετακινήσεων. Ε, επιπλέον, η πρόοδος σε κάποια θέματα σχετίζεται και με την πρόοδο που θα μπορούσε να επιτευχθεί σε άλλα θέματα, ε, κυρίως ε, τον κανονισμό Δουβλίνου και τον κανονισμό για τη διαδικασία ασύλου. Η επόμενη συζήτηση θα γίνει στην ομάδα εργασίας το Μάιο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Η Κομισιόν, μήπως θέλει να πάρει το λόγο. Πολύ σύντομα, ε, αν θέλετε να ευχαριστήσω καταρχάς την εισηγήτρια για το σχέδιο έκθεσης και τις πολύ ενδιαφέρουσε τροπολογίες που υπευλήθησαν. Ε, χαιρόμαστε που το σχέδιο έκθεσης ε, διατηρεί την ισορροπία που προσπάθησε να επιτύχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μεταξύ των στόχων της πρότασης και για να περιορίσουμε τις δευτερογενείς μετακινήσεις και για την ένταξη και την εναρμόνιση των προτύπων και είμαστε βέβαιοι ότι πλέον με τις ε, τροπολογίες θα μπορέσουμε να διατηρήσουμε αυτή την ισορροπία. Επίσης, επισημαίνουμε ότι πολλές από τις τροπολογίες ε, τονίζουν ε, διαδικαστικές εγγυήσεις και μέτρα ένταξης, που είναι άλλωστε και ο στόχος που προσπάθησε να επιτύχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ήθελα επίσης να αναφέρω ότι ανησυχούμε λίγο, διότι αρκετές από τις τροπολογίες σε κάποια μέρη του κειμένου ε, δεν θα μπορούσαν να γίνουν αποδεκτές λόγω της διαδικασίας της αναδιατύπωσης και ε, το διαπιστώνουμε αυτό ε, και γιατί το Συμβούλιο έχει λάβει μια διαφορετική προσέγγιση και ακολουθεί πάρα πολύ στενά τους κανόνες αναδιατύπωσης και το κατά πόσο θα γίνονται παραδεκτές οι τροπολογίες. Αυτά ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ και να δώσουμε τώρα το λόγο στη Σόφη. Ναι, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και να ευχαριστήσω και τους συναδέλφους ε, για τη συνεισφορά τους και για την ε, ευχάριστη συνεργασία που είχαμε στην ομάδα. Ε, να πω λίγα πράγματα. Καταρχάς, αυτό που διέπει εμένα και τη δουλειά μου δεν είναι τόσο ιδεολογία, αλλά να συμπεριφερόμαστε στους ανθρώπους όπως θα θέλαμε να μας συμπεριφέρονται. Επίσης, ε, ε, οι άνθρωποι δεν είναι άγγελοι. Πρέπει να υπάρχουν και ε, κάτι ως δέλεαρ αλλά και ως τιμωρία. Δηλαδή και πρέπει να τους προσφέρουμε και έναν τρόπο ζωής που θεωρούμε εμείς αξιοπρεπή. Και πρέπει να είμαστε ειλικρινείς ε, συνάδελφοι. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή πρόσφυγες οι οποίοι ζουν αυτή τη στιγμή σε συνθήκες που θεωρούμε ότι είναι κάτω των βασικών αναγκών. Ε, σε χειμερινές συνθήκες, για παράδειγμα σε σκηνές, ε, ε, που ούτε καν θα έπρεπε να τις αποκαλούμε σκηνές, στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή το θεωρώ επονίδιστο. Επίσης θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό όχι μόνο σε αυτή την έκθεση αλλά και στην όλη μεταρρύθμιση του συστήματος ασύλου είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν, ε, διότι πιστεύω ακράδαντα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να διαθέτει μια κατάλληλη πολιτική ασύλου για να είναι ανεξάρτητη και από τρίτε χώρε. Έχουμε δει όλοι πόσο δύσκολε ε, έγιναν οι συνθήκε συνεργασία με την Τουρκία και το θεωρώ ε, δυσάρεστο να πρέπει να βασιζόμαστε σε μια τόσο ασταθή και ολοένα και πιο απολυταρχική κυβέρνηση. Θα πρέπει λοιπόν να υποδεχόμαστε αυτούς τους ανθρώπους και να τους επιτρέπουμε να αφομοιωθούν με τον καλύτερο δημετρό τρόπο. Ε, όσον αφορά τα θέματα διεθνούς προστασίας, ε, εγώ συμφωνώ απόλυτα ότι δεν είναι θέμα μετανάστευσης αυτό, οικονομικής μετανάστευσης, αλλά απουσία κατάλληλων οδών για την νόμιμη ε, ε, οικονομική μετανάστευση, οι άνθρωποι θα προσπαθήσουν να καταχραστούν το σύστημα. Ε, δεν μπορούμε να τους κατηγορήσουμε, δεν είναι εγκληματίε γιατί προσπαθούν να βελτιώσουν τον τρόπο ζωής τους, αλλά το σύστημα ασύλου δεν έχει σχεδιαστεί για μετανάστευση για λόγους εργασίας. Γι' αυτό και η πρότασή σας κύριε Πρόεδρε για την μπλε κάρτα είναι πάρα πολύ σημαντική. Πρέπει κατεπηγόντως να έχουμε και ένα σύστημα το οποίο θα παρέχει νόμιμες οδούς για την μετανάστευση παράλληλα με το σύστημα ασύλου. Και επίσης, αυτοί οι άνθρωποι που ε, επικρίνουν αυτούς οι οποίοι ε, καταχρώνται το σύστημα ασύλου είναι αυτοί που δεν θέλουν να μιλήσουν και για τις νόμιμες οδούς μετανάστευσης εργασίας. Δεν μπορούμε να έχουμε ε, δύο μέτρα και δύο σταθμά. Ε, όσον αφορά τις δευτερομεγενείς μετακινήσεις, όλοι συμφωνούμε ότι πρέπει να τις περιορίσουμε και το θέμα είναι αν εδώ θα έχουμε καρότο ή μαστίγιο. Πάντα χρειαζόμαστε και κάποιες τιμωρίες και ο κύριος Αλάχο ε, αναφέρθηκε σε αυτό. Ε, υπάρχουν όμως ε, κυρώσει εδώ. Δεν μπορούν όλοι να κάνουν ό,τι του επιθυμούν και να μην είναι διαθέσιμοι για τις διαδικασίες χωρίς να υπόκεινται τις συνέπειε. Δεν ισχύει αυτό. Υπάρχει περιορισμός ελευθερία, υπάρχει δυνατότητα κράτηση, αλλά θεωρούμε ότι θα πρέπει να είναι λογικά και αναλογικά όλα αυτά τα μέτρα και πρωτίστω αποτελεσματικά. Και βάσει και των πληροφοριών που λαμβάνουμε, Προφανώς και οι δευτερογενείς μετακινήσεις είναι ε, συνέπεια παραγόντων πίεσης. Άνθρωποι που ζουν σε φρικτές συνθήκες κατά πάσα πιθανότητα θα μετακινηθούν σε μια άλλη χώρα. Δεν είναι γιατί θέλουν να πάνε σε μια συγκεκριμένη χώρα, είναι γιατί θέλουν να πάνε κάπου όπου θα μπορούν να ζουν αξιοπρεπώς. Εάν λοιπόν βρίσκονται στο μπάτο σε συνθήκες υποδοχής ε, όσον αφορά ε, κάποιες χώρες, τότε έτσι ενθαρρύνουμε τις δευτερογενείς μετακινήσεις, ακριβώς αυτές που θέλουμε να περιορίσουμε. Όσον αφορά την πρόσβαση στην αγορά εργασία, νομίζω ότι αυτό είναι το πιο περίπλοκο ζήτημα, παρά το γεγονό ότι βλέπω ότι σχεδόν όλε οι πολιτικέ ομάδε έχουν υποβάλει τροπολογίε που περιορίζουν, μειώνουν την περίοδο κατά την οποία δεν υπάρχει καμία πρόσβαση στην αγορά εργασία. Ε, τουλάχιστον λοιπόν συμφωνούμε ω προ την κατεύθυνση που πρέπει να ακολουθήσουμε και καταλαβαίνω και γιατί νιώθουν δυσάρεστα κάποιοι. Ακόμα και στι χώρε όμω όπου υπάρχει αμέσω ή πολύ γρήγορα πρόσβαση στην αγορά εργασία, όπου υπάρχουν Υπάρχουν εκτεταμένα προγράμματα ε, που βοηθούν αυτούς τους ανθρώπους να βρουν μια θέση εργασίας. Τα καλύτερα αποτελέσματα είναι να βρουν το 20% των ετών των άσυλο δουλειά και αυτό στις χώρες που έχουν τα καλύτερα αποτελέσματα. Περί τίνος πρόκειται λοιπόν. Η Ευκαιρίε που έχουν αυτοί οι άνθρωποι να βρουν μια θέση εργασία είναι ελάχιστε, Υπάρχουν τεράστια προσκόμματα. Αυτό που προτείνουμε λοιπόν εμείς είναι να μειώσουμε λίγο κατά αυτά τα εμπόδια και να μεγιστοποιήσουμε αυτές τις ελάχιστες δυνατότητες που έχουμε. Δεν αναφερόμαστε πια και σε μαζική εισρωή ανθρώπων στην αγορά εργασίας ακόμα και αν μπορείτε να επιτύχετε αύξηση κατά 10% ή 15% ε, να βρουν θέση εργασίας αυτοί οι άνθρωποι, ήδη θα είναι πλεονόκτημα. Γιατί ε, ο καθένας θα έχει μια θέση εργασίας, θα είναι εξάρτητος, δεν θα βασίζεται σε κοινωνικά επιδόματα και κατά πάσα πιθανότητα δεν θα μπει και σε μπελάδες. Ε, επομένως, είναι προς το συμφέρον όλων μας να βρουν μια θέση εργασίας αυτοί οι άνθρωποι το συντομότερο δυνατόν. Δύο ακόμα παρατηρήσεις. Πρώτον, θεωρώ ότι μία αρχή την οποία δεν αποφασίσαμε ευθύ εξ αρχής ίσως, αλλά έχω την αίσθηση ότι προκύπτει από τη συζήτηση, η μεταχείριση ε, με τους υπηκόους των χωρών. Ούτε καλύτερα ούτε χειρότερα. Αυτό είναι χρήσιμο. Και επίση θα ήθελα να επισημάνω ότι πρέπει πάντα να έχουμε κατά νου ότι η τελική έκθεση, όπως θα ψηφιστεί στην Ολομέλεια, δεν θα είναι αποτέλεσμα του τριμερούς διαλόγου και παρά το γεγονός ότι υποστηρίζω και συγχαίρω την Μαλτέζικη Προεδρία για την εξαιρετική δουλειά που κάνει, γνωρίζουμε όλοι ότι κάποια κράτη-μέλη θα πιέσουν ε, το Συμβούλιο προς την εντελώς αντίθετη κατεύθυνση. Ε, πρέπει λοιπόν να το έχουμε και αυτό κατά νου. Ε, ψηφίζουμε τις αρχές μας, ε, τα πιστεύω μας, αλλά ξέρουμε και ότι θα ξεκινήσει και η διαπραγμάτευση. Και το Συμβούλιο θα έχει ίσως και μια ακραία θέση. Αυτό το οποίο θα ψηφίσουμε λοιπόν δεν θα είναι το αποτέλεσμα και αυτό πρέπει να το έχουμε κατά νου. Θα γίνει μια ακόμα συνεδρίαση στο Στρασβούργο κατά πάσα πιθανότητα για να ολοκληρώσουμε ε, την έκθεση. Ελπίζω να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε συμφωνία για τις τροπολογίες και να μπορέσουμε να προετοιμάσουμε την ψηφοφορία. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ και την εισηγήτρια και τους σκιώδης εισηγητές γιατί πραγματικά ήταν ε, ε, συζήτηση υψηλού επίπεδου και η ε, νομική βάση είναι άσυλο και μετανάστευση και όχι απασχόληση και γι' αυτό ε, είχαμε σύγκρουση αρμοδιοτήτων με την Επιτροπή Απασχόληση και χρειάστηκε να διαχωρίσουμε τις νομικές βάσεις. Και όπως και εσύ είπε σωστά, υπάρχει αυτή, αυτό το κενό, γιατί δεν υπάρχουν νομοθετικές δίωδοι ε, για ουσιαστική κοινοτική πολιτική που χρησιμοποιεί το κράτη-μέλη και αυτό καθιστά ακόμη πιο περίπλοκο το θέμα. Πάντως νομίζω ότι του αποδώσαμε τη δέουσα προσοχή σήμερα το πρωί και ευχαριστώ θερμά και σένα Σοφή Ιντβέλτ και τους και οδησηγητές γιατί ήταν πραγματικά πολύ διεξοδική συζήτηση και περιστατωμένη. 24-25 Απριλίου θα έχουμε την ε, ψηφοφορία στην Επιτροπή. Και τώρα θα έχουμε μία παρουσίαση, μια και σβήνουν τα φώτα αυτό φαντάζομαι ότι θα έχουμε. Σημείο 17. Όπως ξέρετε, το Φεβρουάριο του 2016 η Ευρωπόλ θέσπισε ένα ειδικό ευρωπαϊκό κέντρο κατά της παράνομης διακίνησης μεταναστών για να αντιμετωπίσει τις οργανωμένες ε, εγκληματικές ομάδες που υποφελούνται από τη λαθροδιακίνηση. Ε, θα έχουμε τώρα την παρουσίαση της ε, έκθεσης δραστηριοτήτων μετά από την πρώτη χρονιά λειτουργίας και καλωσορίζουμε τον επικεφαλής του κέντρου, τον κύριο Κρεπίνκο, το Διευθυντή του Ευρωπαϊκού Κέντρου κατά της παράνομης διακίνησης μεταναστών που θα μας παρουσιάσει, παραλαμβάνω, την έκθεση δραστηριοτήτων των πεπραγμένων μετά την πρώτη χρονιά λειτουργίας. Καλώς ήρθατε κύριε Κρεπίνκο, κύριε Διευθυντά. Περιμένουμε την παρουσίασή σας από το έργο αυτού του Ευρωπαϊκού Κέντρου της Ευρωπόλ για την, κατά της παράνομης διακίνηση μεταναστών. Ε, είναι αυτονόητο ότι νιώθω μεγάλη τιμή που έχω την ευκαιρία να σας παρουσιάσω σήμερα αυτό το πολύ σημαντικό θέμα της έκθεσης ε, πεπραγμένων με, για το τεράστιο καθήκον και σημαντικό καθήκον που έχουμε για την αντιμετώπιση παράνομης διακίνησης μεταναστών κατά δίστακτων ανθρώπων που ε, εκμεταλλεύονται την ευάλωτη κατάσταση πολλών ε, πολιτών για να αποκομίσουν ε, με ανήθικο τρόπο και με σχροκέρδια ωφέλη. Θα σας κάνω μια σύντομη παρουσίαση μικρή του παρελθόντος, του παρόντος και μερικά στοιχεία για το μέλλον. Δεν χρειάζεται να τρέξω σε απόμακρο παρελθόν ξέρετε πώς ε, οι μεταναστευτικές και προσφυγικές ροές έχουν αλλάξει το τοπίο στην Ευρώπη και έχουν ενισχύσει τις κλιματικές δραστηριότητες κάποιων κυκλωμάτων. Γι' αυτό και η Ευρωπόλ χρειάστηκε να προσαρμόσει τις ικανότητές της αλλά και την προσέγγιση της στο φαινόμενο αυτό. Γι' αυτό και πριν από ένα χρόνο εγκαινιάσαμε το Ειδικό Ευρωπαϊκό Κέντρο κατά της παράνομης διακίνησης μεταναστών. Και θα ήθελα να διευκρινίσω ότι μοναδικός μας ε, στόχος είναι να αντιμετωπίσουμε τις ε, οργανωμένες τις συνοριακές εγκληματικές ε, ομάδες που δραστηριοποιούνται σε θέματα παράνομης διακίνησης μεταναστών. Είχαμε λοιπόν πριν από λίγες εβδομάδες την πρώτη μας επέτειο και καλέσαμε ε, τους επικεφαλείς ε, τέτοιων ε, ομάδων, μονάδων, όχι μόνο στα από τα κράτη-μέλη, από και άλλους εταίρους παγκοσμίω. Και εξετάσαμε αυτά τα θέματα και το πώς θα προχωρήσουμε στο μέλλον. Αργότερα θα σας παρουσιάσω τα πεπραγμένα του 2016. Εγώ θα ήθελα να επικεντρωθώ σε κάποια βασικά μας πορίσματα. Συμφωνήσαμε ότι έχουμε ανάγκη όχι μόνο μια διεθνή συνεργασία, αλλά και μια πολυκλαδική διατομιακή συνεργασία, γιατί το θέμα της επιβολής του νόμου αποτελεί μία μόνο πτυχή της αντιμετώπισης αυτού του φαινομένου της ε, παράνομης διακίνησης μεταναστών. Επικεντρωθήκαμε φυσικά στην επιχειρησιακή στήριξη στις ε, έρευνες, ε, και στηριζόμαστε σε κάποιους βασικούς πυλώνες. Θα πρέπει να αντιληφθούμε πώς χρησιμοποιούνται τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για την ε, λαθροδιακίνηση από τους λαθροδιακινητές. Προσπαθούμε να καταλάβουμε, να κατανοήσουμε και να αντιμετωπίσουμε την ε, αύξηση παραχαραγμένων, πλαστογραφημένων εγγράφων ή ταυτοτήτων, αλλά και ακόμη και αυθεντικών που χρησιμοποιούνται για τέτοια λαθροδιακίνηση και προσπαθούμε ε, να δούμε και το φαινόμενο αυτού του σκοτεινού δικτύου του dark web που επίσης χρησιμοποιείται για την παράνομη διακίνηση μεταναστών και μάλιστα εκφράσαμε την ε, ε, στράτευσή μας να αυξήσουμε περαιτέρω την ανταλλαγή πληροφοριών και την κοινή χρήση πληροφοριών, κυρίως για τις τρίτες χώρες, τις εξοκοινωτικές, ιδιαίτερα τις αφρικανικές, γιατί ο διάδρομος της κεντρικής Μεσογείου είναι αυτός που χρησιμοποιείται κυρίως και είναι αντικείμενο κατάχρηση σήμερα από τους ε, παράνομους διακινητές. Για να δούμε τι έκανε η Ευρωπόλ και τα κράτη-μέλη το 2016 από την ε, θέσπιση του κέντρου. Είχαμε μία άνευ προηγουμένου άνοδο του αριθμού των υπόπτων για λαθροδιακίνηση με αναφορέ στη Ευρωπόλ. Πάνω από 17.000 νέοι ύποπτοι προστέθηκαν ε, στη βάση δεδομένων για Έχουμε πάνω από 50.000 συνολικά τέτοιους ελαφροδιακινητές και από, άλλες, ε, από άλλα εγκλήματα έχουμε μετάβαση σε, στη λαθροδιακίνηση γιατί η παράνομη διακίνηση μεταναστών ε, δίνει ευκαιρία για πολύ γρήγορα κέρδη. Και έχουμε ε, εντοπίσει πάνω από χίλιους ύποπτους λογαριασμούς ε, μέσω κοινωνικής δικτύωσης και μαζί με την ε, μονάδα της ε, Ευρωπόλ για το παράνομο περιεχόμενο προσπαθούμε να κατανοήσουμε καλύτερα αυτό το φαινόμενο και να βοηθήσουμε τα κράτη-μέλη να αντιμετωπίσουν και επιγραμμικές ε, δραστηριότητες παράνομης διακίνησης. Δεχτήκαμε γύρω στα 12.000 επιχειρησιακά μηνύματα. Η Ευρωπόλ, όπως ξέρετε, είναι υπεύθυνη μόνο για τα σοβαρά οργανωμένα εγκλήματα με εμπλοκή τουλάχιστον δύο κρατών μέλων Φανταστείτε λοιπόν τι έβρος έχουν αυτές οι δραστηριότητες. Επίσης, ε, πάνω από 2.500 ε, πλαστογραφημένα παραχαραγμένα έγγραφα έχουν ε, καταγγελθεί. Αυτό το θέμα μας απασχολεί ιδιαιτέρως γιατί σήμερα έχουμε την παράνομη διακίνηση αλλά οι συμμορίες ε, που ερευνούμε και που παρέχουν πλαστογραφημένα ή παραχαραγμένα έγγραφα ε, το κάνουν όχι μόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και παγκοσμίω. Και, ε, και άλλε δραστηριότητε οργανωμένου εγκλήματο αξιοποιούν τέτοια πλαστογραφημένα έγγραφα και η τρομοκρατία και όχι μόνο η λαθροδιακίνηση. Είχαμε πάνω από 2.000 νέε υποθέσει πέρυσι. Και επίσης έχουμε διατηρήσει την ισχυρή μα παρουσία και στην Ελλάδα και στην Ιταλία, αλλά και σε χώρες που έχουμε κινητές ομάδες. Πάνω από 1.800 μέρες είχαμε ανάπτυξη προσωπικού μας επιτόπου. Και από κοινού με τους συναδέλφους στη Frontex κάνουμε ενημέρωση των μεταναστών και προσπαθούμε να ακούσουμε τις ιστορίες τους για να κατανοήσουμε καλύτερα τι συμβαίνει ιδιαίτερα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και να αντιληφθούμε πώς λειτουργεί το οργανωμένο έγκλημα, πώς προσελκύει τα θύματα του, να δούμε πώς ε, γίνονται οι πληρωμές και επίσης ακούμε τρόπες ιστορίες για τις ε, συνθήκες ε, διακίνησης, όχι μόνο προς την Ευρωπαϊκή Ένωση από τρίτες χώρες, αλλά και εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εσωτερική διακίνηση μεταναστών. Είχαμε Έχουμε κάθε εβδομάδα, είχαμε κάθε εβδομάδα πέρυσι μια συνάντηση επιχειρησιακού περιεχομένου. Ούτε μια εβδομάδα δεν πέρασε χωρί τέτοια συνεδρίαση, ε, προκειμένου να συνδράμουμε τα κράτη-μέλη να παρακολουθούν τέτοιε υποθέσει ε, και να κάνουμε ένα ακόμη βήμα στην καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματο. Είχαμε 93 ε, υποθέσει υψηλή προτεραιότητα με την πλήρη συνδρομή τη Ευρωπόλ. Μπορεί να μην φαίνεται μεγάλο αριθμό αυτό, αλλά πρόκειται για υποθέσει που εμπλέκουν πολύ περισσότερα κράτη-μέλη, πολύ πάνω από δύο. Και στόχος είναι να διαταράξουμε αυτά τα οργανωμένα κλώματα όσο γίνεται. Όχι μόνο ε, συλλαμβάνοντας ε, λαθροδιακινητές, που είναι η φυσική αυτούργη, αλλά να εντοπίσουμε και τους ηθικού αυτούργου ή του οργανωτές, αυτούς που βρίσκονται στο παρασκήνιο του φαινομένου τη παράνομη διακίνηση. Από ε, αξιωματούχους από τα κράτη-μέλη. Έχουμε αναπτύξει εμπειρογνώμονες μας και στα Ιταλικά κέντρα καταγραφής πρόσφατα, αλλά εδώ και ένα χρόνο και στα Ελληνικά κέντρα καταγραφής και υποδοχής. Όχι μόνο για να εντείνουμε τις ε, δραστηριότητες κατά των λαθροδιακινητών, αλλά και να εξασφαλίσουμε καλύτερους ελέγχους ε, για να αντιμετωπίσουμε κατά πόσο μερικοί τέτοιοι ε, μπορούν να συνιστούν απειλή για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και μάλιστα είχαμε 27 ε, κοινέ ημέρε δράση. Μερικέ ήταν ε, πανευρωπαϊκού χαρακτήρα, οργανώθηκαν πέρυσι από την Ευρωπόλ, με συμμετοχή αστυνομικών αλλά και τελωνιακών και άλλων φορέων, ώστε όχι μόνο να αντιμετωπίσουμε την παράνομη διακίνηση μεταναστών, αλλά και άλλα οργανωμένα εγκλήματα, και να αυξήσουμε τον αντίκτυπό μας σε ομάδες συμμορίες οργανωμένου εγκλήματος. Αυτό ήταν το επιχειρησιακό σκέλος, αλλά υπάρχει και σημαντική στρατηγική πτυχή στο έργο του κέντρου μας. Όχι μόνο η συμβολή μας στο έργο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αλλά και τα Τακτικότητε ενημερώσει προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο. Και αυτά είναι τμήματα της εντολή μα. Έχουμε καθημερινή ενημέρωση των κρατών μελών για το φαινόμενο αυτό, όχι μόνο των κρατών μελών και άλλων βασικών ενδιαφερομένων και έχουμε και στη Γεροπόλη και παγκοσμίω διάφορες εκδηλώσει στι οποίε συμμετέχουμε. Μία αξιοσημεία τέτοια πρωτοβουλία ήταν να αποκοινούμε τη Frontex με συμμετοχούς ε, από την Αφρική έγινε μια τέτοια εκδήλωση στον Νίγηρα ε, προκειμένου να διευρύνουμε τη συνεργασία μας και με ομολόγους μας από την Αφρική. Φυσικά με σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, προστασία των δεδομένων διαπιστώνουμε ότι αν θέλουμε να είμαστε πιο επιτυχεί στην καταπολέμηση και την εξάρθρωση τέτοιων συμμοριών, θα πρέπει να επεκτείνουμε την συνεργασία μας και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ήταν τεράστια επιτυχία που είχαμε στην καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παρ' όλα αυτά, ε, η αντιμετώπιση, εξάρθρωση των συμμοριών εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι πιο δύσκολη. Εκεί υπάρχουν κάποια κενά. Γι' αυτό και χρειαζόμαστε εταίρους και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, για να έχουν και αυτή αποτελεσματική αντιμετώπιση του φαινομένου αυτού. Τώρα λίγα λόγια και για το μέλλον. Σας είπα ποιε είναι οι απόπειρε μα για συνεργασία με βασικέ χώρε τη Αφρικανική Υπήρου. Θα συνεχίσουμε αυτές τις προσπάθειες και τις, ε, τη συνδρομή κινητή με αναλυτές, με εμπειρογνώμονες προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και εκτός Ευρωπαϊκή Ευρωπαϊκής και όπου χρειάζεται φέρουμε τις υπηρεσίες μας κοντά στο πελάτη ώστε να μειώσουμε το χρόνο μετάδοσης των πληροφοριών προς τους άμεσα ενδιαφερόμενους που είναι οι επιτόπου ερευνητές. Επίσης είχαμε την επιχείρηση Σοφία, UNAFROMED και μάλιστα το κέντρο μας εκπροσωπείται και έχουμε καθημερινές ανταλλαγές απόψεων για τις εξελίξεις. Επίσης έχουμε και έξω κοινωτικέ δραστηριότητες, συνεργασία με την Ιντερπόλ στο σχέδιο ISON και άλλα παρεμφερή θέματα. Επίσης έχουμε και μια νέα νομική βάση. Θα έχουμε από την 1η Μαΐου τη νέα νομική βάση με τον νέο κανονισμό της Ευρωπόλ που θα μας επιτρέψει να είμαστε πιο ευέλικτοι στις διεθνείς μας ε, ανταλλαγές. Αλλά φυσικά θα κρατήσουμε το δικό μας στιβαρό καθεστώς προστασίας των δεδομένων που είναι το κλειδί της επιτυχίας της Ευρωπόλ. Κάνουμε ό,τι μπορούμε λοιπόν, βάζουμε τα δυνατά μας για να υλοποιήσουμε ε, τη διακήρυξη της Μάλτας, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στο διάδρομο της Μεσογείου, της Κεντρικής Μεσογείου και φυσικά με συνεργασία με τους εταίρους μας προκειμένου να ενισχύσουμε ε, τις ομάδες επιβολής νόμου και εδώ και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτά είναι συντομία. Ε, πάντως, ποτέ δεν είχαμε τόσες πολλές ε, έρευνες ε, για το δίκτυο, ποτέ δεν είχαμε τόσο εκτεταμένη ανταλλαγή πληροφοριών, ποτέ δεν είχαμε τόσο έντονη στράτευση και δέσμευση για την αντιμετώπιση αυτού του φαινομένου. Παρ' όλα αυτά, μακρύς είναι ο δρόμος που έχουμε ακόμη, γιατί παραλαμβάνω, τα κλώματα αυτά έχουν πλοκάμια και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και σε αυτό το θέμα θα επικεντρωθούμε επίσης στο μέλλον. Αυτά και είμαι στη διάθεσή σας για να απαντήσω στις απορίες σας. Ευχαριστώ κύριε Κρεπίνκο. Είναι πολύ σημαντικό για μας να ενημερωθούμε για τη δραστηριότητά σας κατά την πρώτη χρονιά λειτουργίας σας γιατί είναι σημαντικός ο θεσμικός μας ρόλος στα πλαίσια της λογοδοσίας της Europol. Είναι λοιπόν για μια σειρά από λόγους για τα μέλη μας πολύ σημαντικό. Πολύ σημαντική η λειτουργία του κέντρου σας. Και γι' αυτό δεν θα σας εκπλήξει ότι οι διάφοροι συνάδελφοι θέλουν να πάρουν το λόγο για να σας ε, κάνουν κάποιες ερωτήσεις ή να σχολιάσουν. Ε, όπως σας είπα λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με τον κύριο Ντίαθ Δεμέρα, ο οποίος ε, είναι εισηγητής μας για την Ευρωπόλ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ και τον κύριο Κρεπίνκο για την παρουσία του και για την παρουσίαση ενώπιον της Επιτροπής μας των επιτυχιών, των σαφών επιτυχιών αυτής ε, της ε, πρόσφατης υπηρεσίας που έχει μόνο ένα χρόνο ζωής. Τα αποτελέσματα είναι πολύ θετικά. Λοιπόν, Αναφερθήκατε στις ε, πραγματικές δυνατότητες συνεργασίας με χώρες της Αφρικής και της Μέσης Ανατολής. Αναφερθήκατε στο Νιζέρ, στο Νίγηρα. για να αντιμετωπίσουμε εγκλήματα που έχουν ε, ε, δηλαδή καταστάσεις όπου διαπράττονται πολλά εγκλήματα. Όμως ε, πρόσφατα ο πρώην Γάλλος Υπουργός Εσωτερικών και ο Ισπανός Υπουργός Εσωτερικών πήγαν στον Ήγηρα για να υπογράψουν ένα πρωτόκολλο με την κυβέρνηση της χώρας ακριβώς για την εξουδετερώση των δικτύων. Εσείς έχετε εμπλακεί σε αυτήν την συμφωνία. Αν το EMCS συμμετέχει. EMSC, συγγνώμη. Και κάτι άλλο. Εάν υπάρχουν όντως δυνατότητες ε, ουσιώδης συνεργασίας για την καταπολέμηση του εγκλήματος, ιδιαίτερα στην Αφρική για την καταπολέμηση των ε, δικτύων των ε, εγκληματιών που εκμεταλλεύονται αθώα θύματα. Και νομίζω ότι μπορούμε να... Μπορείτε να μου απαντήσετε χωρίς να θεωρήσουμε ότι είναι εμπιστευτική η πληροφορία. Θα ήθελα λοιπόν να μου πείτε εάν θα μπορούσατε να εγκαταστήσετε κάποιες αντένες προσωπικού στα πιο θερμά σημεία προέλευσης και διαμετακίνησης. Γιατί κατά τη γνώμη μου, άμα θέλουμε να είμαστε αποτελεσματικοί, είναι καλύτερα να μπορούμε να δράσουμε εκεί και όχι μόνο στην Ελλάδα ή την Ιταλία. Όταν ε, φτάσουν τα άτομα αυτά στην Ιταλία, Είμαστε ήδη στο τέλος ε, της ε, διαδικασίας διάπραξης των εγκλημάτων. Εάν μπορούμε να αντιδράσουμε εκεί που ξεκινάει η παραβατικότητα, ίσως μπορούμε να σώσουμε ανθρώπινες ζωές. Και κάτι άλλο. Έχετε στενή σχέση ή έχετε αντιπαράθεση με την Frontex. Βεβαίως καταλαβαίνετε τι εννοώ με αυτή την ερώτηση. γιατί ιδίως ε, στις χερσαίες περιοχές ε, υπάρχει θέμα κοινής αρμοδιότητας. Θα ήθελα να μου πείτε ποιο, ποιος είναι ο διαχωρισμός μεταξύ των αρμοδιοτήτων των δικών σας και της Frontex. Βεβαίως περιμένουμε νέα νομική βάση. Αλλά και αυτή η νέα νομική βάση σχετίζεται με την ημερομηνία της 1ης Μαΐου, οπότε θα έχουμε το νέο κανονισμό για την Ευρω... Ευρωπόλ και θα δούμε τότε πώς ακριβώς θα λειτουργήσουν όλα αυτά. Και σας συγχαίρω για την εργασία σας. Ευχαριστώ. Χρειάστηκε να θέσετε μερικά από αυτά τα θεσμικά θέματα, αλλά παρακαλώ τους συναδέλφους, γιατί έχουμε πολλούς ομιλητές και έχουμε και ψηφοφορίες στις 12. Σας παρακαλώ λοιπόν συνάδελφοι, μήπω θα μπορούσατε να περιοριστείτε σε δύο λεπτά. Ο κύριος Τζούρεκ. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα είμαι σύντομος. Καταρχάς, ευχαριστώ τους προσκεκλημένους για την ε, σκληρή δουλειά που κάνετε. Στόχος μας είναι να υπάρχει ένα πλήρες νομικό πλαίσιο και τώρα να εφαρμοστεί. Οπότε, να θέσω τα εξή ερωτήματα. Πώς θα θέλατε να αλλάξουμε το, το νομοθετικό πλαίσιο για να σας βοηθήσουμε, για να γίνετε πιο αποτελεσματικοί. Υπήρχαν ε, και προηγούμενες προσπάθειες στην Ένωση πριν από δύο χρόνια νομίζω, τον Απρίλιο του 2015 συγκεκριμένα. Το Συμβούλιο της Ευρώπης, μόνο συγγνώμη το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, ε, είπε ορισμένα πράγματα για την ε, τροποποίηση των υποδομών. Αλλά έχουμε τόσα πολλά νομικά εμπόδια και από την άλλη ε, δεν αξιοποιούνται τα μέσα και των, των νομικών μέσων των Ηνωμένων Εθνών γιατί η επιχείρηση Σοφία από ανθρωπιστική άποψη είναι αξιέπαινη, αλλά είναι πολύ περιορισμένη σε εμβέλειας. Επίσης, ε, ίσως θα έπρεπε να οργανωθούμε καλύτερα στο Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. Αλλά η χώρα που φάνηκε να έχει πιο φιλοευρωπαϊκή στάση ήταν το Ηνωμένο Βασίλειο και επ' ευκαιρία θα ήθελα να ευχαριστήσω γιατί έδειξε την καλύτερη στάση υπέρ τη υπεράσπιση των ευρωπαϊκών συμφερόντων στο Συμβούλιο Ασφαλεία του Ηνωμένου Βασίλειου. Η κυρία Ζίπελ. Α, συγγνώμη, Μπρίγκετε. Δεν είσαι ακόμη, δεν είναι ακόμη η σειρά σου. Η κυρία Έρνστ. Κορνέλια, εσύ έχει σειρά. Καλά, δεν θα με πειράζει να μιλήσει η αλλά εντάξει. Κοιτάξτε, αυτό το θέμα με στενοχωρεί λιγάκι. Γιατί η καλύτερη αποτροπή της διακίνησης είναι να υπάρχουν νόμιμοι, νόμιμες οδοί μετανάστευσης. Δεν είναι εδώ λαθρεμπόριο διαμαντιών. Πρόκειται για άτομα που θέλουν να έρθουν στην Ευρώπη από ορισμένε περιοχές. Είμαι ιδιαίτερα λοιπόν ε, αβέβαιοι αν έχουν έννοια αυτά τα πράγματα. Τι δίκτυα είναι αυτά. Ποια δίκτυα καταργήσατε. Εάν ε, διαλυθεί ένα δίκτυο, δεν γίνεται αμέσως ένα άλλο. Οι οποίες κατόπιν ε, θεριεύουν. Πώς λοιπόν αντιμετωπίζετε αυτή την αναγέννησή τους μπορείτε να τη σταματήσετε. Μπορείτε να μας πείτε πιο συγκεκριμένα ποια, πώς ακριβώς ε, λειτουργούν αυτοί οι διακινητές, από πού ξεκινάνε. Θεωρείτε ότι η δραστηριότητά σας όντως ε, τους περιορίζει. Ή μήπως αυξάνεται η δραστηριότητά τους λόγω των συνθήκων στις χώρες προέλευσης. Αυτές προκαλούν, αυτές οι καταστάσεις προκαλούν την δραστηριότητα των διακινητών. Ευχαριστώ. Ο κύριος Στετίνα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ για την παρουσίαση. Πολύ συγκεκριμένη ερώτηση. Σε τι βαθμό η Europol μπορεί να διαλύσει αυτά τα δίκτυα. Να πνίξει αυτή την δραστηριότητα που έχει προκαλέσει αυτές τις ροές από την Κεντρική και Ανατολική Μεσόγειο. Μπορείτε να βοηθήσετε ε, να σταματήσει αυτό. Και πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε εμείς. Η κυρία Κώστα. Ο, ο κύριος Κώστερ. Ευχαριστώ πολύ. Γιατί άτομα. Τι άτομα είναι αυτοί οι διακινητές. Έχουμε διάφορες εκθέσεις ότι εν μέρη είναι άτομα που προηγουμένως ήταν ψαράδες. Και λόγω των ε, εμπορικών συμβάσεων μεταξύ Ένωσης και Αφρικανικών κρατών έχασαν τη δουλειά τους. Μπορείτε να μας πείτε κάτι γι' αυτό. Και ποιοι είναι οι πελάτες τους. Επίσης, για να αντιμετωπίσουμε τη δραστηριότητά τους δεν πρέπει μόνο να δημιουργήσουμε νόμιμες οδούς μετανάστευσης αλλά και να αντιμετωπίσουμε τις συνθήκες που προκαλούν τη μετανάστευση. Ξέρετε πώς αντιμετωπίζουν ακριβώς οι διακινητές τους πρόσφυγες. Τους επιτίθενται το γεγονός λοιπόν ότι τους βάζουν σε βάρκες οι οποίες ε, δεν είναι αξιόπλοες. Δεν σημαίνει αυτό ότι τους υποχρεώνουν, τους επιτίθενται. Δεν ισχύει και αυτό. Ευχαριστώ. Η Body Valor. Χωρίς μικρόφωνο. I'm replacing Jan uh, Αντικαθιστώ το Γιάν σήμερα και μας είπαν ότι όλα τα θέματα της βάσης δεδομένων περιλαμβάνονται εδώ. Συγγνώμη, εγώ το παρέβλεψα πριν ε, συνεχίσεις. Έπρεπε να είχα αναφέρει στην εισαγωγή μου ότι στα πλαίσια της απαλλαγής ε, του προπολογισμού η χρήση των ε, ιδιωτικών βάσεων δεδομένων ε, θα ελεγχθεί και θα έπρεπε να ζητήσουμε πληροφορίες και από αυτού. Έπρεπε να το είχα πει στην εισαγωγή μου και σε ευχαριστώ που το έθιξες. Λοιπόν, το ερώτημα είναι ότι ε, η Ευρωπόλ χρησιμοποιεί ε, μια ιδιωτική βάση δεδομένων και πληρώνει άδεια στην Thomson Reuters κάθε χρόνο. Έχουμε κάποιες ανησυχίες από αυτού, διότι αυτή η βάση δεδομένων είναι αρκετά εμφυλογόμενη πολλές φορές συνδέει ανθρώπους και οργανώσεις με τρομοκρατία μόνο επί τη βάση των δημοσίων ε, πόρων, χωρίς να γίνει έρευνα, να υπάρχει διαφάνεια και να υπάρχουν και αποτελεσματικοί τρόποι αντιμετώπισης. Έχουμε λοιπόν κάποιες ερωτήσεις. Θα θέλαμε να ξέρουμε πώς χρησιμοποιείται αυτή η βάση δεδομένων από την Ευρωπόλη στις καθημερινές εργασίες, αν μπορεί κάποιο ε, να επηρεαστεί επειδή το όνομά του εμφανίζεται στη βάση δεδομένων, ε, πώς διασφαλίζεται ότι οι πληροφορίες είναι σωστές από την Ευρωπόλ, γίνεται κάποια διασταύρωση με άλλες πηγές. Η Ευρωπόλ ισχυρίζεται ότι η χρήση βάσεων δεδομένων όπως η WorldCheck δεν ε, ε, χρησιμοποιείται για να εξετάσουμε την αξιοπιστία της πηγής και την ακρίβεια των πληροφοριών και αν όντως ισχύει αυτό, για ποιο λόγο να τη χρησιμοποιείτε. Και επίσης, ε, πόσο στοιχίζει η άδεια για την βάση δεδομένων WorldCheck κάθε χρόνο και από πότε τη χρησιμοποιείτε. Η Επιτροπή απάντησε σε γραπτό ερώτημα της ε, Σοφή και του Γιάνν ε, πέρσι και είπε ότι κανένας ε, Ευρωπαϊκό Οργανισμό και Υπηρεσία δεν χρησιμοποιεί την βάση δεδομένων αυτή, απάντηση η οποία ήταν ε, ε, ψευδή. Επομένως θα πρέπει να μας δώσετε και ένα επικαιροποιημένο κατάλογο όλων των ευρωπαϊκών οργανισμών και υπηρεσιών που πληρώνουν άδεια για να χρησιμοποιούν αυτή τη βάση δεδομένων. Και όσον αφορά τα, ε, τα θέματα διακίνησης, θεωρώ ότι ο μόνο τρόπο να αντιμετωπίσουμε τους διακινητές είναι νόμιμη οδοί και για τους ετούντες άσυλο αλλά και για τους οικονομικούς μετανάστες. Μόνο έτσι μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τη, αντιμετωπίσουμε τη διακίνηση. Και ως προς τους διακινητές. Ποιοι είναι οι διακινητές. Αυτοί που διακινούν ανθρώπου, Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που βοηθούν και οι εκκλησίες, οργανώσεις κοινωνίας των πολιτών. Αυτοί βοηθούν ανθρώπους. Τους θεωρείτε αυτούς διακινητές. Πού είναι ο ορισμός. Ποια είναι τα όρια του ορισμού. Ίσως θα μπορούσαμε να ρωτήσουμε για τη wall check στη συνέχεια όταν θα απαντήσετε στις υπόλοιπες ερωτήσεις. Η κυρία Βερζιά. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, συγγνώμη έχασα την αρχή της παρέμβασής σας και θα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη. Είμαι εισηγήτρια στην Επιτροπή ε, Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για τα θέματα μετανάστευσης και ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις τρίτες χώρες και θα ήθελα λοιπόν να επικεντρώσω την παρέμβασή μου σε αυτό το ζήτημα. Η συνεργασία με τις χώρες της Αφρικής και μάλιστα στη συνέχεια της εβδομάδας της Μάλτας και με τις χώρες του κέρατος της Αφρικής είναι πολύ σημαντική και σε συνέχεια αυτόν που έλεγε και ο συνάδελφος ε, Διασδεμέρα, η συνεργασία με τι χώρε του κέρατο τη Αφρική δεν θα πρέπει να γίνεται με τι ίδιε συνθήκε και όπω γίνεται με τι χώρε τη Δυτική Αφρική. Ε, τα θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων δεν είναι τα ίδια στην ε, Ανατολική και Δυτική Αφρική, παρά το γεγονό ότι έχουμε να πούμε και άλλα πράγματα για τη Δυτική Αφρική, αλλά υπάρχει μια κάποια διαφορά. Ε, μαζί με κάποιους συναδέλφους ε, και με την ε, συνάδελφο εδώ δίπλα μου, την Κορνίλια, πήγαμε στο Σουδάν το Δεκέμβριο και στη διάρκεια εκείνης της αποστολής ακούσαμε πολλά πράγματα για τη συνεργασία με την Ευρωπόλ. Θα ήθελα λοιπόν να μου πείτε κάποια παραπάνω πράγματα όταν υπάρχει συνεργασία με την αστυνομία μιας χώρας όπως το Σουδάν και λέμε ότι σεβόμαστε τα ανθρώπινα δικαιώματα, θα πρέπει να υπάρχουν και κάποια προληπτικά μέτρα. Δεν είμαι βέβαιη ότι λαμβάνονται αυτά τα μέτρα. Και γνωρίζουμε, παρά το γεγονός ότι δεν ξέρουμε μέχρι ποιο επίπεδο, ε, ότι κάπου συμμετέχουν και οι αρχές του Σουδάν στη διακίνηση ανθρώπων στο Σουδάν. Το Σουδάν είναι ε, πραγματικά κόμβος όσον αφορά τη διακίνηση και έχω κάποιες ανησυχίες ως προς αυτό. Θα ήθελα να σας δώσω ένα παράδειγμα. Εδώ και 9 μήνες ε, τώρα, ένας νέος Ευρωπαίος βρίσκεται στη φυλακή εδώ και 9 μήνες ε, και λέγεται Μπερέ. Είναι από την Ερυθρέα, συγγνώμη και ξέρουν ότι ο άνθρωπος αυτός είναι στο Σουδάν. Ακόμα και αρχές ε, της Ερυθρέας είπαν ότι έγινε λάθος με αυτόν τον άνθρωπο. Οι, οι αρχές του Σουδάν ε, σε θέματα μετανάστευση είπαν ότι πρόκειται περί λάθους και αυτοί. Και παρόλα αυτά αυτό ο νέος άνθρωπος εξακολουθεί να βρίσκεται στη φυλακή. Εάν υπάρχει αστυνομική συνεργασία δεν θα έπρεπε να χρησιμεύει και για τέτοιες περιπτώσεις. Όταν ένας αθώος άνθρωπος βρίσκεται στη φυλακή 9 μήνες λόγω λάθους ταυτότητας ε, δεν θα έπρεπε να γίνει κάτι. Ε, κάτι μου διαφεύγει ποια είναι η πραγματικότητα αυτής της συνεργασίας, ε, σε τι χρησιμεύει και αν δεν χρησιμεύει και στην αθώωση ανθρώπων που βρίσκονται στη φυλακή αδίκως ε, ε, για εννέα μήνες, κάπου κάνουμε κάτι λάθος. Με συγχωρείτε, αλλά αυτή η κατάσταση πραγματικά με ανησυχεί. Ευχαριστώ. Η κυρία Βουίμπερκ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και να ευχαριστήσω και για τις ε, πληροφορίες για την Ευρωπόλ. 50.000 διακινητές. Αδιανόητα υψηλός αριθμός και αντιλαμβάνομαι ότι πολύ δύσκολα μπορούμε να τις παρακολουθήσουμε όλους αυτούς. Η ερώτησή μου είναι η εξής. Όμως ξέρουμε ότι οι μεταναστευτικές ροές από την Τουρκία προς την Ελλάδα μειώθηκαν, αλλά αυξήθηκαν οι ροές από τη Λιβύη προς την Ιταλία. Το Μάρτιο μόνο είχαμε αύξηση κατά 57% σε σχέση με το ίδιο διάστημα πέρσι και αυτό είναι τρομακτικό πολλοί από αυτούς που συμμετέχουν στην έρευνα και διάσωση είναι εθελοντικές οργανώσεις που απλώς προσφέρουν βοήθεια και πλησιάζουν όλο και περισσότερο τις λιβικές ακτές. Το 40% των ανθρώπων που συμμετέχουν σε έρευνα και διάσωση είναι εθελοντικές οργανώσεις. Από τα γερμανικά μέσα άκουσα ότι ο διευθυντής της Frontex επέκρινε το γεγονός ότι αυτές οι εθελοντικέ οργανώσεις συνεργάζονται με τους διακινητές, αλλά θα ήθελα να ξέρω και τη δική σα την άποψη από αυτού. Θεωρείτε ότι αποτελεί πρόβλημα και τι σκοπεύετε να κάνετε. Ευχαριστώ, η Μπεργκή Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, και λυπούμε που παρεξήγησα πριν το νεύμα σα και νόμιζα ότι είχα εγώ σειρά. Είπατε ότι θα πρέπει να κλείσουμε τα κενά στην ανταλλαγή πληροφοριών, βελτιώνοντας αυτή την ανταλλαγή πληροφοριών. Ε, δεν θα ήθελα να ξαναξεκινήσουμε την ενδοευρωπαϊκή συζήτηση για τα προβλήματα που έχουμε στην ανταλλαγή πληροφοριών. Όταν όμως μιλούμε για καταπολέμηση της ε, παράνομης διακίνησης μεταναστών, εκεί πραγματικά θα θέλαμε περισσότερες πληροφορίες για το τι συμβαίνει στις χώρες προέλευσης και διέλευσης. Εξού και η ερώτησή μου είναι αξιόπιστες οι πληροφορίες από τις χώρες αυτές και είναι πρόθυμες οι χώρες προέλευσης ε, να συνεργαστούν με την Ευρωπαϊκή Ένωση και να καταπολεμήσουν πιο αποτελεσματικά το οργανωμένο έγκλημα. Επίσης, όπως είπαν οι συνάδελφοι, είναι σαφές ε, ότι είναι σημαντικές οι αστυνομικέ έρευνε και η συνεργασία με την Ευρωπόλ για να εντοπιστούν αυτά τα εγκληματικά κυκλώματα. Αλλά επίσης είναι σαφές ότι αν επικεντρωθούμε μόνο στην αστυνομική συνεργασία δεν πρόκειται ε, να μας βοηθήσει να λύσουμε το πρόβλημα. Με βάση τις δικές σας ε, πληροφορίες και στοιχεία και τη ενισχυμένη αστυνομική συνεργασία που έχουμε με τρίτες χώρε. Πιστεύετε ότι θα μπορούσαμε να έχουμε συνεργασία και με άλλους φορείς, άλλους οργανισμούς ε, και άλλες διευθύνσεις της Επιτροπής. Ε, για παράδειγμα σε οικονομικά θέματα, αναπτυξιακής βοήθειας και ούτω καθεξής, ώστε να μην επικεντρωθούμε μόνο στην αστυνομική συνεργασία για να καταπολεμήσουμε αυτού του είδους την εγκληματικότητα. Ευχαριστώ. Η Σοφή Ιντφελτ. Μία σύντομη ερώτηση. Όχι για το, την παράνομη διακίνηση μεταναστών, αλλά για τη World Check. Εξεπλάγημα που παρά την αρχική άρνηση ότι χρησιμοποιείται τη World Check, τελικά διαπιστώθηκε ότι και τη χρησιμοποιείται και πληρώνεται ε, τέλη. Και μετά την διαρροή εγγράφων, που δεν ήταν από την Ευρωπόλη διαρροή, ε, αναρωτιέμαι γιατί δεν μας απαντήσατε αμέσως. Γιατί πραγματικά κάτι τέτοιο πλήττει την εμπιστοσύνη μας προς την Ευρωπόλ αν θολώνει τα νερά προς μεθόδους που χρησιμοποιεί. Θέλουμε περισσότερη ενημέρωση για τη χρήση τέτοιων επίμαχων, εμπορικών μάλιστα βάσεων δεδομένων. Στη απάντηση που μας στείλατε είπατε ότι δεν χρησιμοποιείτε την World Check, αυτή τη βάση δεδομένων, για να βρείτε κάποιους, αλλά για να συμπληρώσετε πληροφορίες που ήδη έχετε. Αυτές όμως είναι ε, πληροφορίες από δημόσιες πηγές που δεν ε, ε, έχουν εξακριβωθεί. Πώς χρησιμοποιείτε τέτοιου είδους λοιπόν βάσει δεδομένων ε, και έχετε, ποιες άλλες παρόμοιες βάσεις δεδομένων χρησιμοποιείτε. Όντως, σύνθετες ερωτήσεις, αλλά έχουμε μακρά πείρα με την Ευρωπόλ και κυρίως είναι μια, ένας οργανισμός ε, που συμμετέχει σε ανταλλαγή πληροφοριών ε, και θέματα βάσης δεδομένων και ανταλλαγές προσβάσης σε βάση δεδομένων και το θέμα της παράνομης διακίνησης είναι πολύ σύνθετο, πολύ πλευρό ε, και οι αρμοδιότητες είναι πολλαπλές, το είπε και ο κύριος Δίας Δεμέρα. Θα ήθελα παρακαλώ να μου απαντήσετε. Ευχαριστώ και ευχαριστώ πραγματικά για το μακροσκελή κατάλογο ερωτήσεων που μου υποβάλλετε και τα πολύ άριθμα σας σχόλια. Θα κάνω ό,τι μπορώ για να απαντήσω σε όλες τις απορίες. Θα ήθελα όμως πρώτα να επισημάνω κάποια στοιχεία. Ξέρω ότι γνωρίζετε την Ευρωπόλ, την εντολή της και τον τρόπο που εμείς λειτουργούμε στα πλαίσια αυτά. Θα ήθελα να τονίσω ότι όλες οι πληροφορίες της βάσης δεδομένων μας στέλνονται στη, στο κέντρο μας από τα κράτη-μέλη. Και όχι μόνο από τα κράτη-μέλη, αλλά και από τους επιχειρησιακούς μας εταίρους και από άλλους οργανισμούς που δεν έχουν κατά σχέση με την επιβολή του νόμου. Ο Σιμών θα μιλήσει αργότερα για το συγκεκριμένο θέμα της βάσης δεδομένων World Check. Ίσως δεν ήμουν αρκετά σαφή στην εισαγωγή μου, αλλά σε ό,τι αφορά τη συνεργασία με την Αφρική και τις αφρικανικές χώρες, προς το παρόν είναι μηδενική αυτή η συνεργασία. Η Ευρωπόλ δεν έχει άμεσες σχέσεις με οποιαδήποτε αρχή επιβολή νόμου σε οποιαδήποτε αφρικανική χώρα. Είμαστε υπερήφανοι για το έργο που επιτελούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και γνωρίζουμε ότι από τη στιγμή που έχουν φτάσει στην ευρωπαϊκή επικράτεια οι λαθροδιακινητές και οι μετανάστες. Είναι πολύ δύσκολο ε, να εμποδίσουμε τις δραστηριότητες τους. Ε, αλλά το, αυτό είναι το δεύτερο σκέλος της δραστηριότητας. Το πρώτο είναι πώς ξεκινάει η παράνομη διακίνηση. Γι' αυτό θέλουμε συνεργασία, είπαμε, ε, με τις άλλες αφρικανικές χώρες. Αλλά υπάρχουν προβλήματα και προς την προς τον έλεγχο των δεδομένων, την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ούτω καθεξής. Γι' αυτό και είμαστε πολύ προσεκτικοί και η πρόοδος είναι πολύ αργή με τις αφρικανικές χώρες. Πάντως, εμείς παρουσιάσαμε το έργο της Ευρωπόλ και τις ευκαιρίες που περιέχει και από τις 25 χώρες που συμμετείχαν στον Ήγηρα στο σεμινάριο εκείνο, λίγες ήρθαν και εκδήλωσαν ενδιαφέρον για πιθανή συνεργασία στο μέλλον. Ε, βρισκόμαστε ακόμη στα σπάργανα αυτή της διαδικασίας ε, που θα είναι αρκετά χρονοβόρα. Και ως προς την πρώτη σας ερώτηση. Ε, είχα συναντήσει με εμπειρογνώμονες από την Ισπανία και τη Γαλλία που ήταν παρόντες στον Ήγυρο και στην κοινή επιχειρησιακή μονάδα με τις αρχές του Νίγηρα και της Νιγηρίας και τους είπα ότι και η Ευρωπόλ θα υποφεληθεί από την έκβαση αυτής της συνεργασίας που όπως σας, είπα βρίσκεται σε πολύ προκαταρκτική φάση. Και αυτό θα είναι και το μοντέλο που θα χρησιμοποιήσουμε και στο μέλλον. Δηλαδή, ένα κράτος μέλος ε, επιτόπου θα λαμβάνει πληροφορίες από μυστικές υπηρεσίες και θα είναι ο θεματοφύλακας αυτών των πληροφοριών ε, με πλήρη σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των άλλων πτυχών και μετά το κράτος μέλος θα ε, διαβιβάσει αυτά τα στοιχεία στην Ευρωπόλ ώστε να ε, πληρώσουμε αυτά τα κενά στην πληροφόρηση και να συνδέσουμε κάποιες πιθανές υποθέσεις στην Ευρώπη με αντίστοιχε στην Αφρικανική. Προς το παρόν λοιπόν δεν έχουμε σχηματίσει ε, πείρα από την συνεργασία με την Αφρική. Τώρα ξεκινά και θέλουμε να μπει στα σκαριά και να βελτιωθεί. Και προσπαθούμε να έχουμε κάποιες πληροφορίες και από τα ε, βασικά κέντρα της Αφρικής, τους κόμβους, να δούμε ποια είναι τα κίνητρα ε, για τους πρόσφυγες να προσφύγουν σε τέτοια κυκλώματα λαθροδιακινητών, πώς λειτουργούν και να δούμε και τους κινδύνους στους οποίους εκτίθενται αυτοί οι άνθρωποι. Επίσης, να δούμε πώς τους προσελκύουν οι λαθροδιακινητές. Όλοι γνωρίζουμε ότι ε, η οικονομική, η δινή οικονομική κατάσταση στις αφρικανικές χώρες είναι ένα κίνητρο και η μεταφορά στην Ευρώπη είναι μια απόδειξη επιτυχίας ε, όταν κάποιος καταφέρνει και φτάνει στην Ευρώπη και μπορεί να στέλνει λεφτά πίσω στην οικογένειά του. Οπότε δεν είναι μυστήριο ποιο είναι το κίνητρο, αλλά είναι τρομακτικό ε, πόσο πληρώνουν στους λαθροδιακινητές τι χρέη κάνουν προκειμένου να πληρώσουν τους ελαφροδιακινητές και επίσης σε τι κινδύνους εκτίθενται. Και για τις επιχειρήσεις ε, έρευνας και διάσωσης δεν είναι δική μας αρμοδιότητα. Πάντως, άσχετα με το πόσο κοντά στις λιβικές ακτές ε, γίνονται αυτές οι επιχειρήσεις, παρόλα αυτά έχουμε, είχαμε άνευ προηγουμένο μεγάλο αριθμό πνιγμών στη Μεσόγειο. Και φαντάζομαι δυστυχώς θα συνεχιστεί αυτό η κατάσταση. Σε ό,τι αφορά τη Frontex, μετά την ενίσχυση της εντολής και των ικανοτήτων θα μας βοηθήσει και η Frontex με επιπλέον πληροφορίες από, τη, από τις συνοριακές περιοχές και τη διασυνοριακή εγκληματικότητα. Η Europol θα είναι ο βασικός οργανισμός συγκέντρωσης πληροφοριών και εμείς θα, στη, θα συνδράμουμε με πληροφορίες για σοβαρό και οργανωμένο έγκλημα και πολλές από τις ε, πληροφορίες που λαμβάνουμε στα σύνορα μπορεί να ενδιαφέρουν μία συγκεκριμένη χώρα, να μην ε, συμπληρώνουν τη συνολική κατάσταση, αλλά ίσως και αυτέ οι πληροφορίες οι ε, βοηθήσουν. Τώρα, σε ό,τι αφορά τη νομική βάση, η νέα νομική βάση θα μας επιτρέψει να διευρύνουμε τις σχέση μας με τρίτες χώρες που δεν έχουν συνάψει συμφωνία σύνδεση με την Ευρωπόλ, οπότε έχουμε μία διεύρυνση εκεί και θα έχουμε ε, την ευκαιρία να συνεργαστούμε και με άλλους τομείς που δεν αφορούν μόνο την επιβολή του νόμου. Βέβαια δεν θέλουμε να διευρύνουμε υπερβολικά το φάσμα, γιατί είμαστε ένας οργανισμός που συνδράμει κυρίως ε, τα κράτη-μέλη στην καταπολέμηση του σοβαρού και οργανωμένου εγκλήματος. Υπάρχουν λοιπόν αρκετές δυνατότητες, αλλά θέλουμε να διαφυλάξουμε το στιβαρό καθεστώς που έχουμε ε, για τα δεδομένα και την ασφάλεια των πληροφοριών μας. Σε ό,τι αφορά τα δίκτυα αυτά, τα κυκλώματα και πώς οργανώνονται, ε, πριν από μία εβδομάδα δημοσιεύσαμε την ΣΟΚΤΑ, την ε, μελέτη απειλών τέτοιων δικτύων, που δεν είναι μόνο ε, δίκτυα παράνομης διακίνησης, αλλά γενικώ ε, σοβαρού οργανωμένου εγκλήματος στην Ευρώπη και εκτός Ευρώπης. Πάνω από 5.000 τέτοιες εγκληματικές συμμορίες εντοπίσαμε στην Ευρωπαϊκή Επικράτεια, που παίρνουν διάφορες μορφές οργανωμένου εγκλήματος. Έχουμε τις πιο παραδοσιακούς τρόπους οργανωμένου εγκλήματος, όπου έχουμε έναν αρχηγό και μια πολύ ιεραρχική δομή, ε, άκαμπτη. Με ίσως ε, και οικογενειακούς δεσμούς, ε, εθνικότητα, ειδικότητε, αλλά έχουμε και πιο χαλαρά δίκτυα, μικρές ομάδες που συνεργάζονται για τη διάπραξη περιορισμένων εγκληματικών δραστηριοτήτων. Διαφορετικές οι λοιπόν. Και κάτι τέτοιο α, αντανακλά την, τον την καθημερινότητά μας και αυτή τη χαλάρωση που διαπιστώνεται και στους επιχειρηματικούς δεσμούς, στους οικονομικούς δεσμούς, ψάχνουμε να βρούμε το πιο φθηνό τρόπο μεταφοράς, ε, να βρούμε τα πιο φθηνά ή τα πιο προσιτά πλαστογραφημένα έγγραφα. Αυτά για τους διακινητές. Και είναι δύσκολο να βρούμε έναν ελάχιστο κοινό Πάνω από 100 εθνικότητες μπλέκονται και μεγάλη πλειοψηφία των κυκλωμάτων που έχουν εξαρ... εξαρθρωθεί ήταν ε, από πολλές ε, εθνικότητες, ακόμη και από πολλές θρησκευτικέ ομάδες. Και παρόλα αυτά αυτοί οι άνθρωποι συνεργάζονται εύκολα παρά τη διαφορά στη θρησκεία ή στην εθνικότητα. Δεν έχουμε μια συγκεκριμένη μορφή ενός κυκλώματος ή μιας ε, εγκληματικής συμμορίας δικτύου. Είναι πολλές οι μορφές. Τώρα, πώς προσπαθούμε να παρεμποδίσουμε τις δραστηριότητες τους ε, στη διόδο της κεντρικής Μεσογείου, σας το εξήγησα προηγουμένως. Και έχουμε έναν ε, ε, εκπρόσωπο από την επιχείρηση Σοφία που συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό Κέντρο κατά της παράνομης διακίνησης ε, μεταναστών και βλέπουμε πώς ε, γίνεται αντιληπτή η επιχείρηση Σοφία επιτόπου, ποια είναι τα αποτελέσματά της. Και φυσικά το βασικό μας ατού είναι οι πληροφορίες που συγκεντρώνουμε και με τις οποίες τροφοδοτούμε και τα υπόλοιπα κράτη-μέλη, όχι μόνο την Ιταλία και την Ελλάδα, για να τα βοηθήσουμε να καταπολεμήσουν αυτά τα κυκλώματα παράνομης διακίνησης. Με ρωτήσατε και για τους διακινητές στην Αφρική. Δεν έχω απάντηση, γιατί όπως είπα και προηγουμένως δεν έχει ξεκινήσει ακόμη συνεργασία. Τώρα αρχίζει και σκιαγραφείται αχνά η μορφή που θα λάβει η συνεργασία μας με τις αφρικανικές χώρες αλλά ακόμη δεν έχει πάρει τέτοια έκταση ώστε να μπορώ να σας ενημερώσω για αυτά αποτελέσματα. Ελπίζω στο μέλλον ε, να έχουμε περισσότερες πληροφορίες, όχι μόνο από ε, αφρικανικές χώρες, αλλά και από άλλους φορείς. Τώρα, ε, η μετανάστευση είναι ένα πολυσύνθετο περίπλοκο φαινόμενο και σίγουρα η συνεργασία με τις αρχές επιβολής του νόμου δεν θα είναι πανάκια. Και μία από τη, είναι μία από τις δραστηριότητες, ένα μακρύ κατάλογο δραστηριοτήτων. Συμμετείχα στην ε, συνεδρίαση των ε, υψηλόβαθμων αξιωματούχων ε, στη Βαλέτα μετά την διάσκεψη κορυφής της Βαλέτα πριν από λίγες εβδομάδες και εκεί εξετάσαμε πέντε πυλώνες για την αντιμετώπιση της μετανάστευσης. Φυσικά θα πρέπει να δούμε τα αίτια τα βασικά και σίγουρα η επιβολή του νόμου είναι ένα από τα εργαλεία της εργαλειοθήκης μας, αλλά όχι το μοναδικό. Και σίγουρα όχι κάποιο μαγικό θαυματουργό εργαλείο. Τώρα, αν μπορούμε να ορίσουμε τους διακινητές. Η Ευρωπόλ δεν ορίζει την έννοια του διακινητή, του λαθροδιακινητή. Μιλούμε για υπόπτους παράνομης διακίνησης μεταναστών. Υπόπτους που έχουν εντοπίσει τα κράτη-μέλη. Πρόκειται για ύποπτο σε μία ποινική έρευνα στα κράτη-μέλη και ενημερώνεται η Ευρωπόλ ε, και ειδοποιείται ότι ο ΤΑΔΕ θεωρείται ύποπτος για παράνομη διακίνηση. Υπάρχουν μικροδιαφορές, αλλά όχι ιδιαίτερες διαφορές ό,τι αφορά τον ορισμό της παράνομης διακίνησης. Διευκόλυση ε, λάθρο μετανάστευσης ή παράτυπης ή παράνομης μετανάστευσης. Ε, υπάρχουν μικροδιαφορές στον ορισμό και ο ορισμός γίνεται από τα κράτη-μέλη, όχι από την Ευρωπόλ. Επίσης, συμφωνώ ότι υπάρχει μια τεράστια διαφορά μεταξύ του κέρατος της Αφρικής και της Δυτικής Αφρικής. Και όπως είπα, αυτό θα το δούμε περισσότερο στο μέλλον. Έχοντας φυσικά πάντα κατά νου ε, τα ανθρώπινα δικαιώματα, την προστασία των δεδομένων και ούτω καθεξής. Εμείς δεν μπορούμε να επηρεάσουμε τις δραστηριότητες ε, των αφρικανικών χωρών, Επίσης θα ήθελα να αποσαφηνήσω ότι η επιβολή του νόμου σημαίνει επιβολή του εθνικού δικαίου, αλλά έχουμε την υποχρέωση να εξασφαλίζουμε και την τήρηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων κατά την εφαρμογή του νόμου. Νομίζω ότι απάντησα σε όλες τις ερωτήσεις και αν ε, μου διέφυγε κάποια, ζητώ συγγνώμη, αλλά πολύ ευχαριστώ να απαντήσω και στις υπόλοιπε αν υπάρχουν. Η κυρία Βερζιά, έχω την εντύπωση ότι προσπαθήσατε να απαντήσετε στην ερώτησή μου, αλλά ίσως δεν ήμουν αρκετά ακριβή ή υπήρχε κάποιο πρόβλημα. Αυτά τα οποία μας είπαν επιτόπου και οι αρχές του ΣΥΔΑΝ και οι αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιτόπου, υπάρχει συνεργασία της Ευρωπόλ με την αστυνομία του Σουδάν και αν ναι, ε, σε ποια φύση, γιατί δεν είναι πράγματα τα οποία μάθαμε στους διαδρόμους, μας τα είπαν οι αρχές του Σουδάν και οι εκπρόσωποι της πρεσβείας μας εκεί επιτόπου και η αποστολή μας που μας είπαν ότι υπάρχει τέτοια συνεργασία. Τι συνεργασία λοιπόν υπάρχει μεταξύ Σουδάν και Ευρωπόλ. Δεν θα ήθελα να σχολιάσω τις πηγές σας ή τι σας είπαν. Είμαι βέβαιος ότι αυτό που σας είπαν, ε, σας το είπαν καλή την πίστη, αλλά η Ευρωπόλη δεν έχει συνεργασία με τις αρχές του Σουδάν. Εντάξει. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Κρυπίνκο, και ευχαριστώ και την ομάδα σας. Τρεπίνκο. Και όπως βλέπετε υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον ε, και επομένως θα θέλαμε να έχουμε συνεργασία σε διοργανικό επίπεδο, σε οποιοδήποτε επίπεδο. Και θα ήθελα να το εκλάβετε αυτό ως ένδειξη του ενδιαφέροντός μας για τη δουλειά σας. Ε, υπάρχουν βεβαίως τεχνικές πτυχές, αλλά υπάρχουν και πτυχές ανθρωπίνων δικαιωμάτων που μας απασχολούν. Και ελπίζουμε φεύγοντας από εδώ να γνωρίζετε ότι εμείς σκοπεύουμε να συνεχίσουμε. Ε, να ενδιαφερόμαστε για τα θέματα αυτά. Ε, θέλετε να μιλήσετε κι εσείς. Ζητώ συγγνώμη. Πρέπει να απαντήσετε και το θέμα της Walser που νομίζω ότι είστε υποχρεωμένοι βεβαίως ε, η Σόφη είναι έχει και άλλη δουλειά γιατί γι' αυτό και είχα και εγώ το μυαλό μου ε, αλλού. Σόφη, προσέχεις εδώ για την απάντηση. Κύριε Πρόεδρε, αξιότυπα μέλη, ε, ευχαριστούμε που ζητάτε από την Ευρωπόλ να σας δώσει περαιτέρω πληροφορίες για τη βάση δεδομένων Wallcheck. Ο ο ρόλος της Ευρωπόλ είναι να βοηθήσει την Ευρωπαϊκή Ένωση στην καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος και της τρομοκρατίας όπως καθορίζεται στην ε, νομική βάση. Και ε, διεκπεραιώνουμε πληροφορίες και επεξεργαζόμαστε πληροφορίες επί τη βάση ε, ε, διαδικασιών που ξεκινούν τα κράτη-μέλη και επιχειρησιακοί εταίροι. Τα όσα κάνουν λοιπόν ε, οι εταίροι ε, διασταυρώνονται με τις βάσεις δεδομένων της Ευρωπόλ. Όπως ξέρετε εφαρμόζουμε υψηλά πρότυπα για να αξιολογήσουμε την αξιοπιστία των πηγών ε, και την ακρίβεια των πληροφοριών που παρέχονται από τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τους επιχειρησιακούς εταίρους μας και τα κριτήρια έχουν καθοριστεί επισήμως στο άρθρο 29 του νέου κανονισμού της Ευρωπόλ αξιολόγηση της αξιοπιστίας των πηγών και ακρίβειας των πληροφοριών. Είναι νομική απέτηση και πάντα εφαρμόζονται αυτά τα πράγματα από την Ευρωπόλ στην πράξη. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε ότι βάσει του άρθρου 29 στο οποίο αναφέρθηκα, η αξιολόγηση συγκεκριμένων δεδομένων και πληροφοριών από την Ευρωπόλ γίνεται κάθε μήνα ε, με τα κράτη-μέλη που παρέχουν τις πληροφορίες. Η World Check ε, δίνει συγκεκριμένες πληροφορίες ανοιχτής ε, πηγής, ε, όπως και άλλα εργαλεία λοιπόν είναι διαθέσιμα στην Ευρωπόλ για να συμπληρώσουν πληροφορίες που είναι ήδη διαθέσιμες, κάτι το οποίο είναι πάγια πρακτική και στα κράτη-μέλη. Οι πληροφορίες από ανοιχτέ πηγές όπως η Walls ε, ε, Check δεν χρησιμοποιούνται για να ε, διαπιστώσουμε την αξιοπιστία των ε, πηγών και την ακρίβεια των πληροφοριών ε, που διατίθενται από τις χώρες μέλη και τους εταίρους μας για επιχειρησιακά θέματα. Επιτρέψτε μου τώρα να σας δώσω κάποιες πιο πρακτικές λεπτομέρειες. Χρησιμοποιούμε πάντα ανοιχτές πηγές για να συμπληρώσουμε πληροφορίες, αλλά ποτέ για να τις αξιολογήσουμε. Επειδή είμαστε ένας Κόμβο πληροφοριών, και αυτό είναι βασικά καθήκοντα της Ευρωπόλ, σκοπεύουμε να ε, ε, προσέχουμε διάφορες πηγές πληροφορίες. Ε, τίποτα δεν ξεκινάει για θέματα επιβολής του νόμου, έρευνα κλπ. επί τη βάση ανοιχτών πηγών. Προσπαθούμε απλώς να λάβουμε περιττέρω πληροφορίες για να συμπληρώσουμε την εικόνα που έχει διαμορφωθεί σε εθνικό επίπεδο. Ε, και όταν χρησιμοποιούμε τέτοιε πηγέ ε, το υποδεικνύουμε στα κράτη-μέλη. Γιατί χρησιμοποιούμε τη WellCheck. Είναι ένα σύνολο αξιόπιστων ανοιχτών πηγών, ε, έχουν δικαστικέ αποφάσει και πολλά άλλα πράγματα. Σε ασφαλέ περιβάλλον μπορούμε να διασταυρώσουμε πληροφορίε που έχουμε από τις εθνικές αρχές με πληροφορίε που λαμβάνουμε από αυτέ τι ανοιχτέ πηγέ. Είναι πάγια πρακτική πλέον να αναζητούμε στο διαδίκτυο πληροφορίε για υπόπτουν αλλά ποτέ δεν δίνουμε μεγαλύτερη σημασία σε αυτές τις πληροφορίες από ό,τι θα έπρεπε να έχουν. Η wall check μας επιτρέπει να το κάνουμε γρήγορα, με ενοποιημένο τρόπο, χωρίς να πρέπει να διατρέξουμε χιλιάδες ιστοσελίδες με μη ασφαλή τρόπο. Γίνεται με διαφάνεια, γιατί η wall check βρίσκεται στον κατάλογο των συμβάσεων της Europol και είναι προσβάσιμο στην ιστοσελίδα μας. Νομίζω ότι αυτό απαντά και στο βασικό θέμα, στο, για το πώς και πότε χρησιμοποιούμε τη World check. Και να σας ε, απαντήσω γραπτός ε, στα πιο συγκεκριμένα ερωτήματα από πότε και πόσο στοιχίζει, γιατί εγώ είμαι στις επιχειρήσεις, δεν είμαι στις προμήθειες. Ναι, νομίζω ότι θα ήταν ε, χρήσιμη και για την Μπόντιλ και για τη Σοφία μια γραπτή απάντηση. Σας παρακαλώ να συμπεριλάβετε και αυτά τα οποία μόλις μας είπατε στην γραπτή σας απάντηση. επειδή κάποιοι συνάδελφοι που έκαναν την αρχική ερώτηση δεν είναι παρόντες. Σας παρακαλώ να αποστείλετε λοιπόν μια γραπτή απάντηση στη γραμματεία μας. Σας ευχαριστώ πολύ συνάδελφοι για την αναλυτική συζήτηση. Ευχαριστώ για την παρουσίασή σας. Λοιπόν τώρα να περάσουμε στο σημείο 18. Πρόταση για τροπημένη οδηγία για την μπλε κάρτα, συνθήκες ε, εισόδου και παραμονής ε, υπηκόων τρίτων χωρών ε, με υψηλό επίπεδο ειδίκευσης. Είχαμε 509 τροπολογίες από αυτού. Έγιναν μια σειρά συνεδριάσεις των σκιωδών. Τους ευχαριστώ πάρα πολύ για την πολλή δουλειά και την αφοσίωσή τους στο θέμα αυτό να σας περιγράψω ποια είναι η κατάσταση όσον αφορά τις προτάσεις μου λοιπόν για συμβιβαστικές λύσεις, για βασικά θέματα και μετά θα ακούσουμε τη γνώμη των σκιωδών. Καταρχάς, όσοι συνάδελφοι δεν έχουν ασχοληθεί με το θέμα αυτό, η συνολική μου προσέγγιση είναι να διασφαλίσουμε επειδή δεν αξιοποιείται πάρα πολύ, επειδή δεν έχουμε πολλά μέσα νόμιμης μετανάστευσης, όπως είπαμε στο προηγούμενο θέμα, δεν έχουμε πολλές δυνατότητες και δεν αξιοποιούμε και αυτή που έχουμε αρκετά. Και κυρίως αξιοποιείται σε μία ή δύο χώρες, αλλά ακόμη και εκεί όχι ιδιαίτερα. Στόχος μας λοιπόν είναι μέσω της αναθεώρησης του συστήματος της μπλε κάρτας να αυξήσουμε την αξιοπιστία του, να μπορεί να αξιοποιείται. Πότε θες το λόγο, Νεταλή? Εντάξει, σημειώνω. Λοιπόν, αυτή είναι η γενική μου στάση. Ευχαριστώ τους Σκιώδης για την εργασία τους για το θέμα αυτό. Είπα λοιπόν 509 τροπολογίες και θέλω να εξηγήσω και, σε όλους τους άλλους συναδέλφους ε, συνεργαζόμεθα με βάση το άρθρο 54 με την, ε, με την Επιτροπή Απασχόλησης. και η Jean Lambert ε, είναι η συγγήτρια και είναι θετικό ότι είναι ενεργό μέλος και της Επιτροπής μας για τα θέματα που έχουν να κάνουν για τα κριτήρια εισδοχής, άρνησης και απόσυρσης και πρόσβασης στην αγορά εργασίας, που το συζητήσαμε και προηγουμένως. Η Επιτροπή λοιπόν Απασχόλησης έχει πλήρη αρμοδιότητα για τα θέματα αυτά. Θα έχουμε λοιπόν πολύ ενδιαφέρουσα συνεργασία με την Επιτροπή Απασχόλησης. Πού βρισκόμαστε. Έχουμε 509 τροπολογίες για τα εξής κυρίως θέματα. θέματα τα θέματα των ε, εθνικών προγραμμάτων σε αντιπαράθεση με ένα ενωσιακό πρόγραμμα όπως είναι η μπλε κάρτα. Ορισμένες άλλες τροπολογίες ε, προτείνουν να συνεχιστούν παράλληλα με το σύστημα της μπλε κάρτας τα εθνικά συστήματα. Αλλά όπως γνωρίζουν οπωσδήποτε και οι σκιώδεις, δεν υπέβαλα τροπολογίες σε αυτό το τμήμα της πρότασης. Και επειδή δεν υπάρχει πολύ προσοχή στο σύστημα αυτό και δεν υπάρχουν αρκετές, μάλλον ελάχιστες μπλε κάρτες δίνονται με βάση αυτό το σύστημα, εμείς πιστεύω πρέπει να στηρίξουμε ένα σύστημα που θα ε, ενθαρρύνει περισσότερο τα κράτη-μέλη να αξιοποιήσουν αυτό το σύστημα, γιατί αλλιώ η αναθεώρηση θα είναι σε επίπτωση. Η μετανάστευση, όπως ξέρετε, είναι πολύ ευαίσθητο θέμα, πρώτο θέμα στα πρωτοσέλιδα είναι μία από τις λίγες δυνατότητες νόμιμης μετανάστευσης. Πρέπει λοιπόν να διασφαλίσουμε να έχει έστω ένα αποδεκτά υψηλό επίπεδο χρήσης. Ορισμένα άλλα θέματα όπου θα υπάρξουν συμβαστικές τροπολογίες. Έχουμε τα θέματα των ορισμών, 27 τροπολογίες για διάφορα θέματα του άρθρου 2 που αναφέρεται στους ορισμούς. Για διάφορα στοιχεία τι σημαίνει υψηλού επίπεδου ειδίκευσης και τι σημαίνει ε, εκπαίδευση ανώτατου επίπεδου και τι σημαίνει υψηλές επαγγελματικές δεξιότητες και τι ακριβώς είναι η επιχειρηματική δραστηριότητα και αν θα έπρεπε να υπάρχει ένας καθορισμένος κατάλογος ή ανοιχτός κατάλογος ε, δραστηριοτήτων που μπορούν να θεωρηθούν επαγγελματικές. Θα υποβάλω λοιπόν συμβαστικές τροπολογίες για το θέμα αυτό των ορισμών. Άλλο βασικό θέμα πεδίο εφαρμογή της μπλε κάρτας. 28 τροπολογίες. Όπου ορισμένοι λένε να επεκταθεί το πεδίο εφαρμογή για να συμπεριλάβει και όσους δεν έλαβαν ε, διεθνή προστασία, κάτοικοι, συγγνώμη, πήκοοι τρίτων χωρών και άλλοι θέλουν να περιοριστεί το πεδίο εφαρμογής. Θα προτείνω ένα συμβαστικό λοιπόν συμβασμό και εδώ. Άλλο θέμα. Πολύ λεπτό αλλά για διαφορετικούς λόγους. Το θέμα των κατοφλίων αποδοχών. Πολλές τροπολογίες. Άρθρο 5. Ορισμένοι λένε ότι πρέπει να παλιφθεί, άλλοι λένε να διατηρηθεί ως υποχρεωτικό και άλλοι λένε να αλλάξει το πεδίο εφαρμογή των ε, κατοφλίων αυτών. Είναι λεπτό θέμα κοινή αρμοδιότητα με την Επιτροπή απασχόληση, Είναι προτεραιότητα και για μένα και για όλους τους κοιόδης. Θέλουμε να επιτύχουμε ένα συμβιβασμό και στις δύο επιτροπές για το θέμα αυτό. Σίγουρα οι σκιώδεις το συζήτησαν. Λεπτό θέμα, βασικό θέμα. Και μεικτή αρμοδιότητα με την ε, Επιτροπή Απασχόλησης. ο ε, μακροπρόθεσμος χαρακτήρας της κινητικότητας, μακροπρόθεσμη κινητικότητα. Και τέλος, ε, τι θα γίνει με την οικογενειακή επανένωση, εάν κάποιος λάβει μπλε κάρτα. Και εδώ θα προτείνω έναν ε, συμβιβασμό για να ανταποκριθώ σε μια σειρά από που αφορούν την πρόσβαση στην αγορά εργασία των μελών τη οικογένειας, τα δικαιώματά τους στα πλαίσια της μακροπρόθεσμης κινητικότητας των κατόχων μπλε κάρτας. Όλα αυτά τα θέματα τα συζητάμε και με τους σκιώδες της ΛΥΜΠΕ και με τους σκιώδες της ΕΜΠΛΕ. Νομίζω ότι έχουμε καλή μέθοδο συνεργασίας με την ΕΜΠΛ, αλλά βέβαια περιπλέκει το θέμα. γιατί από τη μία έχουμε την νομική βάση για τη μετανάστευση και από την άλλη την νομική βάση για την αγορά εργασίας. Η προσέγγιση μου λοιπόν θα είναι να γίνει πιο ορατό, πιο χρήσιμο αυτό το σύστημα της μπλε κάρτας. Καταλαβαίνω ότι υπάρχουν πολλές ευαισθησίες για το θέμα αυτό. Αυτή τη στιγμή δεν πολύ δουλεύει. Θέλουμε λοιπόν κάπως ε, να το βελτιώσουμε. Σας περιέγραψα τις λεπτομέρειες που χρειάζεται να εξεταστούν. Ευχαριστώ τους Κιώδης και τώρα να δώσω το λόγο στους συναδέλφους. Οι συντονιστές ε, ΕΛΚ και ECR δεν είναι παρόντες, οπότε την Ναταλή Γκρισμπέκ που είναι συντονίστρια της ΑΛΔΕ. Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν, σε ευχαριστώ για τη φιλόδοξη έκθεσή σου. Που, όπως είπες, ε, μιλά για την ευελιξία του μηχανισμού της πλε κάρτας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, προσπαθώντας να την καταστήσει πιο ελκυστική. Κάτι που είναι καλή βάση των εργασιών μας επί της οδηγίας αυτής, που η ομάδα μου θεωρεί ε, ως πολύ χρήσιμο εργαλείο για να γίνει πιο ελκυστική η Ευρώπη ως χώρος απασχόλησης. Και σε ευχαριστώ γιατί δεν αποκλείσει κανένα τη συνεργασία. Επιδεικνύεις αυτό το γνωστό βρετανικό fair play και είσαι πολύ διαλλακτικός στις συναντήσεις, πολύ πρόθυμος να βρούμε συμβαστικές λύσεις γιατί είναι η πλειάδα οι ε, τροπολογίες, γύρω στους 600 δεν θυμάμαι καλά. Η ομάδα μου ξεκινά από τη δική σου διαπίστωση ότι η Ευρωπαϊκή Οδηγία για την μπλε κάρτα που έχει εγκριθεί πριν από μία δεκαετία περίπου δεν λειτουργεί αρκετά καλά ή καθόλου μερικές φορές καλά. Και το αποτέλεσμα είναι ότι ελάχιστη είναι κάτοχη τη μπλε κάρτα. Οπότε ελάχιστα αξιοποιείται η οδηγία. Άλλωστε συνοδεύεται από τέτοια γραφειοκρατία και τόσο ε, επαχθείς ε, διατυπώσεις που αποθαρρύνει του επίδοξου ε, δικαιούχους. Οπότε είναι κάπω απεσιόδοξη αυτή η διαπίστωση, αλλά καθιστά αναγκαία την ε, αλλαγή. Άλλωστε και τα κράτη-μέλη μερικές φορές δεν προώθησαν, δεν διαφήμισαν δεόντως ή δεν ενθάρρυναν ε, κάποιους να χρησιμοποιήσουν αυτό το εργαλείο, την μπλε κάρτα, για να προσελκύσουν ε, ταλέντα με υψηλέ δεξιότητε στην Ευρώπη. Οπότε έμεινε αναξιοποίητη η οδηγία. Η Άλντε είναι υπέρ της ε, ενίσχυσης της ευελιξίας, κάτι που φαίνεται και από τις τροπολογίες μας. Θέλουμε απλούστευση των διαδικασιών των προθεσμιών και των διατυπώσεων ε, και μια μεγαλύτερη ευελιξία τους και θεωρώ ότι πολύ εύστοχα αντιμετωπίσει αυτό το θέμα. Επίσης θέλουμε να διευρύνουμε την μπλε κάρτα σε περισσότερους δικαιούχους. Τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει ότι θα πρέπει να δούμε και το θέμα του κατώτατου ορίου μισθού που αναφέρει η οδηγία. Γιατί με βάση τις αναλύσεις και τις εκθέσεις ε, που έγιναν σε ό,τι αφορά την, ε, την έλλειψη λειτουργίας της οδηγίας, θεωρεί ότι το κατόφλι είναι βασικό στοιχείο. γιατί η έλλειψη του κατοφλίου δεν κάνει καθόλου ελκυστική την μπλε κάρτα και εμποδίζει όσους έχουν χαμηλούς μισθούς να ζητήσουν την μπλε κάρτα, μια και δεν τους εξασφαλίζει κάτι καλύτερο. Οπότε ας μην περιορίσουμε την μπλε κάρτα μόνο σε κάποιους με υψηλές δεξιότητες, γιατί χρειαζόμαστε και άλλες δεξιότητες που μπορεί να μην εμπίπτουν στο, στην έννοια της υψηλής ειδίκευσης. Και σε κάποιους τομείς θα πρέπει να προσαρμόσουμε την οδηγία στην πραγματικότητα της εκάστοτε αγορά εργασίας. Αυτά ως προς το δύο. Φαντάζομαι θα το επεξεργαστείτε περαιτέρω, ώστε να καταλήξουμε σε κάποιες συμβαστικές προτάσεις. Και τέλος, ένα κέριο σημείο κατά τη γνώμη μου, θέλουμε ενδεχομένως ένα σύστημα που θα είναι μακροπρόθεσμα πανευρωπαϊκό. Εξού και στις τροπολογίες μας προτείναμε ένα μεταβατικό καθεστώς, πολιετές, ώστε κάποια στιγμή σταδιακά να έχουμε ως απότερο στόχο μια ευρωπαϊκή μπλε κάρτα που θα αντικαθιστά τα εθνικά συστήματα ή τα ανταγωνιστικά συστήματα. Έτσι θα έχουμε ένα διαφανέστερο σύστημα πιο αποτελεσματικό, πανευρωπαϊκής εμβέλειας ώστε να είμαστε πραγματικά ανταγωνιστικοί στην Αμερικανική πράσινη κάρτα ή την Καναδέζικη αντίστοιχη, την Αυστραλέζικη αντίστοιχη πράσινη κάρτα, ώστε να γίνει η Ήπειρός μας ελκυστική ως χώρος απασχόλησης, κάτι που θα ανταποκρίνεται στους ε, ε, στόχους που διατρανώνουμε στις διάφορες συζητήσεις μας. Ευχαριστώ, Νατάλη. Η Μπάρμπαρα Σπινέλη από την ΚΟΕ. Θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την εξαιρετική συνεργασία με όλους εμάς ε, τους και οδησίγητες και να πω ότι εγώ ξεκίνησα από την προϋπόθεση ότι η μπλε κάρτα που δημιουργήθηκε το 2009 ήταν αποτυχία από πολλές κοπιές. Μόνο μια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης τη χρησιμοποίησε με σημαντικό τρόπο, η Γερμανία, και όχι γιατί η Γερμανία είναι πιο Ευρωπαία από άλλες χώρες, αλλά γιατί η κάρτα δεν λειτουργεί ως έχει και υπάρχουν χώρες που έχουν κριτήρια εισδοχής πολύ καλύτερα και ε, πιο ε, ε, επικεντρωμένα στην ένταξη, όπως η ιδέα. Οι περισσότερες τροπολογίες μας, λοιπόν, είναι ε, για να βελτιώσουμε την μπλε κάρτα και να φροντίσουμε τουλάχιστον αυτή η νόμιμη οδός μετανάστευσης να λειτουργεί και να έχει την ισχύ που έχει η Αμερικάνικη πράσινη κάρτα. Γι' αυτό ακριβώ, όπως και ο εισηγητής, πρότεινα και οι αιτούντες άσυλο να μπορούν να κάνουν αίτηση για μπλε κάρτα και θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό η επαγγελματική εμπειρία τριών ετών του μετανάστη να αναγνωρίζεται ε, ως αντίστοιχη πανεπιστημιακού τίτλου σπουδών. Επίσης με τις τροπολογίες μου θα ήθελα να διαγράψω ή να περιορίσω τα πιο σημαντικά για την, τα πιο σημαντικά εμπόδια για την απόκτηση της κάρτας, το πολύ υψηλό όριο ε, μισθού, το οποίο ήταν μέχρι τώρα ένας από τους βασικούς παράγοντες για τη μη λειτουργία της κάρτας και προτείνω επίσης να περιορίσουμε βάζοντας σαφείς ε, όρους τη δυνατότητα των κροατών να διακόψουν προσωρινά την πρόσβαση στην αγορά εργασίας ε, στους κατόχους ε, μπλε κάρτας. Επιπλέον, έχω συμπεριλάβει στις προτάσεις μου και τη δυνατότητα να κάνει κάποιος αίτηση για μπλε κάρτα διαδικτυακά. Επίσης, όπως και ο εισηγητής, ε, έχω συμπεριλάβει αρκετά πράγματα για τη διευκόλυνση της ευρωπαϊκής κυκλοφορίας και την επανένωση με την οικογένειά τους. Επίσης, ε, με χαρά διαπιστώνω ότι αρκετοί από τους κοιόδης εισηγητές έκαναν αντίστοιχες τροπολογίες με τις δικές μου και ελπίζω ότι θα συμφωνήσουμε και θα έχουμε μια έκθεση ε, στο μέτρο του δυνατού φιλόδοξη. καλή επιτυχία λοιπόν στον εισηγητή. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, Μπάρμπαρα. Η Μπόντουν, πριν αρχίσω, επειδή έγιναν πολλές αναφορές στο σουηδικό σύστημα, θα ήθελα να πω ότι χαίρομαι που ετέθη το θέμα αυτό από την Μπόντουλ, διότι σίγουρα πρόκειται για καλό πρόγραμμα και θα μας το εξηγήσετε σίγουρα τώρα στην παρέμβασή σας πώς ακριβώς λειτουργεί. Ε, είναι και η σκιώδη για τους πρασίνους άλλωστε. Ευχαριστώ πολύ. Πράγματι, συχνά αναφέρομαι στο σύστημα της Σουηδίας, γιατί πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ καλό. Έγινε μια μεγάλη αλλαγή πριν από κάποια χρόνια και πρόκειται για μια αλλαγή που οδήγησε σε πολύ θετικά αποτελέσματα και γι' αυτό και το αναφέρω πολύ συχνά. Θεωρώ ότι είναι καλό το γεγονός ότι εξετάζουμε την οδηγία αυτή για άτομα υψηλής εξειδίκευσης είναι καλύτερη βάση, επιτρέπει καλύτερη κινητικότητα και νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας έκανε μια αρκετά καλή πρόταση, αλλά εμείς εδώ από πλευράς Κοινοβουλίου μπορούμε να τη βελτιώσουμε περαιτέρω. Το πρόβλημα το οποίο διαπιστώνω είναι ότι στην Ευρώπη πρέπει να μπορούμε να προσελκύσουμε ε, γενικότερα περισσότερη μετανάστευση για λόγους εργασίας. Εδώ αναφερόμαστε σε άτομα υψηλή ειδίκευση και πριν ήμασταν πολύ αυστηροί επ' αυτού. Στη Σουηδία εκδόθηκαν 8 μπλε κάρτε αν δεν κάνω λάθος, αλλά ταυτόχρονα υπήρχε μεγάλη εισρωή μεταναστών ανθρώπων υψηλής ειδίκευση για πολλά χρόνια, ε, οι οποίοι ήρθαν βάσει του εθνικού μας συστήματο. Βάσει τις οδηγίες θα μπορούσαμε να ε, δυσκολέψουμε αυτούς τους ανθρώπους, αλλά και άλλους, να έρθουν στην Ευρώπη ε, για το σουηδικό σύστημα. Αλλά τώρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έθεσε το εξής ε, ερώτημα θα μπορούσαμε να έχουμε εθνικά συστήματα τα οποία θα λειτουργούσαν εκ παραλλήλου με την οδηγία. Πρέπει να σκεφτούμε επίσης ότι ο πληθυσμός στην Ευρώπη γυράσκει. Η μόνη Ήπειρος που δεν έχει αυτή τη στιγμή ε, πληθυσμό που γυράσκει είναι η Αφρική. Δεν ξέρω τι γίνεται με τη Μέση Ανατολή, αλλά πριν από μερικά χρόνια έτσι είχαν τα πράγματα. Δεν έχω τώρα στατιστικά στοιχεία για τη Μέση Ανατολή. Πέραν της Αφρικής όμως, Υπάρχουν ε, γυράσκουσες κοινωνίες σε όλες τις υπόλοιπες υπήρους, επομένως όλοι ε, θα στραφούν στη συνέχεια σε αυτούς τους πόρους. Πρέπει λοιπόν να μπορέσουμε να προσελκύσουμε όχι μόνο τους ε, ανθρώπους υψηλής εκειδήγευσης, αλλά και τους υπόλοιπους. Στη Σουηδία ε, δεν είχαμε σε κάποια φάση μετανάστευση για λόγους εργασίας. Όλοι περνούσαν από το σύστημα ασύλου και αυτό οδήγησε σε σχεδόν κατάρρευση του συστήματος ασύλου. Οι περισσότεροι εκμεταλλεύτηκαν το σύστημα ασύλου για να λάβουν άδεια εργασία. Όταν άλλαξε η νομοθεσία και επιτρέψαμε και σε άτομα υψηλή ειδίκευση αλλά και σε άτομα χαμηλότερη ειδίκευση να μπορούν να κάνουν αίτηση για άδεια εργασία. μειώθηκαν οι πιέσει ε, από το σύστημα ασύλου και αυτοί που έρχονται πλέον μπορούν να κάνουν αίτηση για άδεια εργασίας πριν ε, φτάσουν στη Σουηδία. Δημιουργήσαμε λοιπόν ένα νόμιμο τρόπο για μετανάστευση για λόγους εργασίας για όλες τις κατηγορίες. Γεγονός το οποίο μας επέτρεψε να βάλουμε τάξη στο σύστημα ασύλου. Οι ετούντες άσυλο περνούν από το σύστημα σύλλου και οι οικονομικοί μετανάστες, όπως τους αποκαλούμε πλέον, ε, ακολουθούν την άλλη οδό. Την μετανάστευση για λόγους εργασίας. Και μετά είχαμε την κατάσταση που ε, ανέφερα προηγουμένως. Κάποιοι από τους οποίους έρχονται ως ετούντος άσυλο θεωρούν ότι έχουν ε, δικαίωμα ασύλου, αλλά λόγω των αυστηρών κανόνων που έχουμε για το άσυλο αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη, απορρίπτεται η αίτησή τους. Αυτοί που έχουν εργαστεί για κάποιο διάστημα στη Σουηδία έχουν ε, τη δυνατότητα να συνεχίσουν ε, την παραμονή τους ως μετανάστες εργαζόμενοι. Το σύστημα αυτό έχει αποτελέσματα. Υπήρχαν κάποια προβλήματα στην αρχή με τους μισθούς και κάποια άλλα. Ε, προσπαθούμε να τα επιλύσουμε και οι εταίροι μας από την αγορά εργασίας συμμετέχουν πολύ. Ε, τα συνδικάτα μας εξηγούν αν κάποια πράγματα δεν έχουν αποτέλεσμα, αν είναι πολύ χαμηλή μισθή. Ε, εμείς πιστεύουμε ότι θα πρέπει να δίνεται αντίστοιχος μισθός για αντίστοιχη εργασία. Ε, και όσον αφορά τα ε, όρια στην οδηγία έχουμε αντίστοιχη προσέγγιση. Εμείς δεν έχουμε όρια, έχουμε διαπραγματεύσεις μεταξύ της αγοράς εργασίας για το τι ισχύει σε κάποια συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία. Αν εγώ είμαι κυπουρός με πολλά προσόντα, θα πρέπει να λαμβάνω τον ίδιο μισθό με έναν ε, ε, Σουηδό επαγγελματία κυπουρό. Πρέπει λοιπόν να έχουμε ένα σύστημα το οποίο λειτουργεί αποτελεσματικά σε όλες τις χώρες. Όσον αφορά αυτό στο οποίο αναφέρθηκε η Μπάρμπαρα. Δυνατότητα ε, για αίτηση για μπλε κάρτα σε αιτούντες άσυλο. Υπάρχει μεγάλος αριθμός ε, αιτούντων άσυλο με υψηλή εξειδίκευση αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη, οι οποίοι απλώς περιμένουν την έκδοση της απόφασης. Κάθονται ε, μπορεί να έχουμε χειρουργούς για παράδειγμα, ο οποίος περιμένει απλώς, έχει όλα αυτά τα προσόντα και τις δεξιότητες, αλλά δεν του επιτρέπεται να εργαστεί και ε, μπορεί να μην τον χρειάζονται μέσα στη Σουηδία, αλλά μπορεί να είναι απαραίτητο στη Γαλλία. Είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν αυτά τα άτομα υψηλής εξειδίκευσης να μπορούν να κυκλοφορούν μέσα στην Ευρώπη ε, εν αναμονή της έκδοσης απόφασής τους για το άσυλο. Ε, ξέρω ότι αυτή η ιδέα θα φανεί ε, παρατραβηγμένη σε κάποιους γιατί υπάρχουν διαφορετικά συστήματα ασύλου σε κάθε χώρα αλλά γνωρίζω ότι υπάρχει και μια περιέργεια για το τι ακριβώς κάναμε εμείς στη Σουηδία και πώς τα καταφέραμε και αναρωτιούνται και αρκετές χώρες πώς θα μπορούσαν να αλλάξουν τα δικά τους τα συστήματα εδώ πρόκειται περί οικονομικών μεταναστών. Δεν είναι άτομα μόνο υψηλή εξειδίκευση, αλλά θα υπάρξει και μεγάλη εισρωή άλλων οικονομικών μεταναστών και δεν θα σταματήσουν να έρχονται απλώς και μόνο ε, επειδή θα σταματήσει ο πόλεμος ε, στη Συρία θα συνεχιστούν αυτές οι ροές ε, και ε, συνεχίζεται εδώ και χρόνια και δεν έχουμε βρει ένα σύστημα ε, για τους ανθρώπους χαμηλής εξαντιδίκευσης. Ή θα πάνε από, την, το διάβλο του ασύλου ή θα έρθουν παράνομα στη χώρα και θα ελπίζουν να μην τους εντοπίσουν και θα δουλεύουν παρανόμως αντί να δουλεύουν νομίμως και να πληρώνουν και φόρους. Νομίζω λοιπόν ότι είναι καλύτερο η οδηγία αυτή να ξεκινήσει, να λειτουργεί, να γίνει μια πολύ καλή ε, συζήτηση. Έχουμε και το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή εδώ. Θα ήθελα να ακούσουμε και τις δικές τους τις σκέψεις. Ε, τι άλλο θα μπορούσαμε να έχουμε για το θέμα αυτό και πώς μπορούμε να κάνουμε τα πράγματα κάπως διαφορετικά. Σας ευχαριστώ. Κατάλαβα, Μποντήλ, ότι σε ενδιαφέρει πολύ αυτό το θέμα. Ναι, σε παρακολουθούσα το αντίστοιχο θέμα όταν έγινε η σχετική μεταρρύθμιση στη Σουηδία. Ναι, έκανα το γνωστό βρετανικό χιούμορ. Εν πάση περιπτώσει. Η κυρία Γκάμπριλ ήταν η σκιώδη γιατρή από το ΕΛΚ, ο Ιωσδόφσκι από το ECR, Φεράρα και Λεμπρετών από το ΙΕΝΕΦ. Ε, ε, δεν μπόρεσαν να παρευρεθούν, αλλά παρακολουθούν το θέμα. Και αυτό και η Κριστίν. Ευχαριστώ. Θα ήθελα και εγώ να σε ευχαριστήσω γιατί είναι πολύ σημαντικό και αξιόλογο το έργο σας σε αυτό το θέμα. Συμφωνώ ότι η μεταρρύθμιση της οδηγίας, η αναθεώρηση της οδηγίας θα πρέπει να μας επιτρέψει να ενισχύσουμε τους νόμους διάβλους πρόσβασης και να καταστήσουμε την μπλε κάρτα πιο ελκυστική και μάλιστα σε όλα τα κράτη-μέλη. Θα ήθελα να σταθώ σε δύο τροπολογίες που κατέθεσα. Την 148 που αφορά την ανάγκη διεύρυνση της πρόσβασης στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Υπηρεσιών Απασχόλησης, το ΕΡΕΣ, και σε πολίτες τρίτο χωρών, σε υπηκός τρίτο χωρών, γιατί το ΕΡΕΣ συγκεντρώνει τις προσφορές απασχόλησης στην Ευρώπη. Ε, η ελκυστικότητα της μπλε κάρτας θα εξαρτηθεί από τη δυνατότητα υπηκών τρίτων χωρών να βρουν εύκολα μια θέση εργασίας στην Ευρώπη. Θα πρέπει να μπορούν να έχουν πρόσβαση στην ολόκληρη την αλυσίδα για την αναζήτηση θέση απασχόληση, οπουδήποτε στην Ευρώπη. Επίση, η τροπολογία 151 αφορά τη διεύρυνση τη κάρτα, τη μπλε κάρτα στο να καλύπτει το σύνολο των εργαζομένων, γιατί θα παραμείνει ελλειπέ το εργαλείο αν ε, επικεντρώνεται μόνο στους εργαζομένους υψηλή ειδίκευση. Θέλουμε να καλύψουμε όλες τις ειδικότητε, ε, όλες τις δεξιότητε όπου λείπουν ε, εργατικά χέρια, όχι μόνο περιορισμό στην υψηλή ειδίκευση. Γιατί έτσι θα ανταποκριθούμε και στις σημαντικές δημογραφικές προκλήσεις με τον γυράσκοντα πληθυσμό μας γιατί έχουμε και θα έχουμε όλο και περισσότερο ανάγκη εργατικό δυναμικό. Θέλουμε λοιπόν ένα ισορροπημένο σύστημα ε, μπλε κάρτες ε, ισοδύναμου, σε όλους τους ε, απασχολούμενους, όλους τους εργαζόμενους στην Ευρώπη και όχι μόνο σε μια κατηγορία τους υψηλά ειδικευμένου. Όπως είπε η Μποντήλ, έχουμε εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Δεν ξέρω να, θα θέλετε να προσθέσετε κάτι. Ε, έγιναν εκτενεί συζητήσει και τέθηκαν ερωτήσεις για την ανάγκη διεύρυνση του πεδίου εφαρμογή για να προσελκύσουμε και άλλους ε, μετανάστες ε, με δεξιότητες και όχι μόνο τους υψηλή ειδίκευση. Αυτό είναι θέμα προσυζήτηση. Καταρχήν, ας εφαρμόσουμε καλύτερα ε, τους ε, υφισταμένους διάβλους που έχουμε και σε εθνικό και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, γιατί δεν έχουμε εναρμόνιση και καλύπτουν τους ανειδίκευτους ή τους χαμηλής ειδίκευσης εργαζόμενους. Υπάρχουν τέτοιες ευκαιρίες, δεν αξιοποιούνται όμως. Επίσης, ε, να συζητήσουμε και περαιτέρω το θέμα περισσότερων κανόνων, γιατί τώρα έχουμε τον έλεγχο καταλληλότητας των κανόνων για την νόμη μετανάστευση και ίσως χρειαστούμε και περισσότερους κανόνες για τους χαμηλής και μέση δίκευσης. Πάντω όταν μιλούμε για την μπλε κάρτα, μην ξεχνάτε ποιο είναι ο στόχο αυτής της οδηγίας, που είναι η βελτίωση των κανόνων στο να προσελκύσουμε υψηλή ειδίκευση εργαζομένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αν διαβρύνουμε υπερβολικά το πεδίο εφαρμογή αυτή τη συγκεκριμένη οδηγία, τότε θα χάσουμε την ευκαιρία να βελτιώσουμε τι σχετικέ διατάξει και να καταστήσουμε πραγματικά ελκυστικότερη αυτή την μπλε κάρτα, γιατί θα δίνουμε περισσότερα δικαιώματα ε, και να στους κατόχους τους, ε, της μπλε κάρτας είναι γιατί μιλούμε για συγκεκριμένη κατηγορία εργαζομένων που θέλουμε να προσελκύσουμε. Και το ίδιο ισχύει για τα κράτη-μέλη. Οπότε αυτή τη στιγμή θα πρέπει να επικεντρωθούμε στη βελτίωση του συγκεκριμένου εργαλείου. Και είμαι ευγνώμων ε, προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο γιατί υποστηρίζει τους στόχους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Μπορεί να υπάρχει κάποια διάσταση σε επιμέρους θέματα, αλλά γενικώ το Κοινοβούλιο είναι υπέρ της πρότασης. Αλλά μην αποσπά η προσοχή μας σε άλλα θέματα, γιατί το θέμα είναι η εργαζόμενη υψηλή δίκευση. Επίσης, ε, θέλουμε νόμιμους διάβλους για τους επικούς και για την νόμιμη μετανάστευση και για άλλους λόγους. Νόμιμη μετανάστευση, συγγνώμη, και για άλλους λόγους. Ναι, ναι, καταλάβαμε, καταλάβαμε ποιο είναι το αντικείμενο. Το επανέλαβες αρκετές φορές. Απλώς ε, ήθελα να ενημερωθούν και οι υπόλοιποι συνάδελφοι γιατί οι σκιώδεις ε, ε, εισηγητές είναι εξοικειωμένοι. Πάντως σας ευχαριστώ θερμά για το ενδιαφέρον που δείχνετε. Φαίνεται και από την πληθώρα τροπολογιών. Θα καταρτήσω τις συμβεστικές τροπολογίες το συντομότερο δυνατό, ώστε να ψηφίσουμε στην Επιτροπή μας στις, 30, στις 3 συγγνώμη, Μαΐου. Εντάξει, πολύ ωραία. Α, ωραία, έχουμε και περιθώριο για ένα 20 λεπτό διάλειμμα, γιατί στις 12 θα ξεκινήσουν οι ψηφοφορίες. Αλλά να είστε στην αίθουσα 12 παρα 5, γιατί θα με μαλώσουν αν δεν αρχίσω ο τις α, ε, ψηφοφορίες, ιδιαίτερα ημέρα 5. Ευτυχώς που είμαστε κοντά στην καφετερία, οπότε να είστε πίσω παρακαλώ 12 παρα 5.

Καθίστε παρακαλώ συνάδελφοι. Θα ξεκινήσουμε αμέσως. Okay, colleagues, um, Λοιπόν, συνάδελφοι. Καταρχήν έχετε όλοι, ελπίζω, τις ηλεκτρονικές κάρτες ψηφοφορίας. Και αν κάποιος την ξέχασε, να το δηλώσει παρακαλώ. Ωραία όλοι. Τις έχετε φέρει. Για την σειρά των σημείων που θα ψηφίσουμε... Δεν υπάρχει πρόβλημα. Ξεκινάμε το πρώτο θέμα ε, για την ασπίδα προστασίας και τελευταίο θέμα θα είναι έκθεση γραπίνη. Δύο ανακοινώσει καταρχήν ε, για το πρώτο θέμα της ασπίδας προστασίας για την ιδιωτικότητα. Κύριε Μπροκ, τι γίνεται, έχετε την κάρτα σας. I'm just, I mean, these are close votes. I want to make sure everyone is settled and... Παρακαλώ, καθίστε όλοι. Μην βιάζετε και τραυματιστείτε με την ησυχία σας. Εντάξει, βολευτήκατε όλοι. Έρχεται και η κυρία Στίβενς. Ένα μόνο ξέχασε την ηλεκτρονική κάρτα ψηφοφορίας. Επειδή ίσως είναι οριακές ε, οι διαφορές, η γραμματεία θα σημειώνει την ψήφο του. Αν κάποιος άλλος ξέχασε την κάρτα να το πει, για να το λαμβάνουμε υπόψη. Η Άλντε ζήτησε ονομαστική ψηφοφορία για την τελική ψηφοφορία στο ψήφισμα για την ασπίδα προστασία ε, για την ιδιωτικότητα. Με βάση τον, το άρθρο 248 παράγραφος 3, και το 68α, 20% των μελών της Επιτροπής θα πρέπει να συμφωνήσει με το αίτημα της ονομαστικής ψηφοφορίας, δηλαδή 12 ευρωβουλευτές θα πρέπει να συμφωνήσουν. Νομίζω ότι έχουμε αυτή την πλειοψηφία. Έχουμε κάποιες προφορικές τροπολογίες, την 5, Weidenholzer 10, Χόλτζερ 35, Ιντερ 46, Λέναρτ Holmeyer 59 Ernst. Το γνωρίζετε ότι είναι προφορικές αυτές οι τροπολογίες. Είπα ποιες θα είναι για να ξέρετε. Δεν θα διαβάσω το περιεχόμενο, να ξέρετε ότι αυτές που σας διάβασα οι τροπολογίες θα είναι προφορικές. Θα διαβαστούν κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας, ως συνήθως. Ξεκινάμε. Τροπολογία 6, άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Παρακαλώ το ΕΛΚ να συνεννοηθεί. Ο κύριος Σόγκορ έχει χάσει την κάρτα του. Ο κύριος Μπρόκ την ξέχασε, θα ψηφίζει με το χέρι. Όταν είναι αρνητικό το δάχτυλο, όταν αντίχειρα προς τα κάτω, έλεγες προς τα πάνω. Να ξέρουν οι συνάδελφοι τι θα ψηφίζουν. Απορρίπτεται. Τροπολογία 9. Άρχεται η ψηφοφορία. Όχι, λάθος λέει ο πρόεδρος. Τροπολογία 7 πρώτα. Άρχεται η ψηφοφορία. Καλά, έχετε δίκιο που φωνάζετε. Εγώ έκανα λάθος. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται τροπολογια 9 Άρχιτε ψηφοφορια Απορρίπτεται. Τροπολογία 10. Προφορική τροπολογία για την αφαίρεση του αποκλειστικό και μόνο, το Σόλουμπι. Άρχιτε ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 11. Άρχεται ψηφοφορία. Τέλος. Εγκρίνεται. Τροπολογία 12. Άρχεται ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 13. Άρχεται ψηφοφορία. Τέλος. Απορρίπτεται. Τροπολογία 14. Έναρξη ψηφοφορίας. Τέλος. Απορρίπτεται. Τροπολογία 15. Έναρξη ψηφοφορία. Τέλος. Εγκρίνεται. Τροπολογία 16. Άρχεται ψηφοφορία. Τέλος. Εγκρίνεται. Τροπολογία 19. άρχιτη ψηφοφορία. Τέλος. Απορρίπτεται. Τροπολογία 20. άρχιτη ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 22. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος. Εγκρίνεται. 23. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος. Εγκρίνεται. Τροπολογία 25. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος. Εγκρίνεται. 26. Άρχεται ψηφοφορία. Τέλος. Απορρίπτεται. 27. Άρχεται ψηφοφορία. Τέλος. Εγκρίνεται. 28. Άρχεται ψηφοφορία. Τέλος. Εγκρίνεται. 29. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος. Απορρίπτεται. Τροπολογία 30. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος. Απορρίπτεται. Α, συγγνώμη, εγκρίνεται. 32. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος. Απορρίπτεται. Τροπολογία 31. Άρχεται ψηφοφορία. Τέλος. Εγκρίνεται. Τροπολογία 43. Άρχεται ψηφοφορία. Τέλος. Εγκρίνεται. Τροπολογία 38. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος, εγκρίνεται. 34. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος. Εγκρίνεται. Τροπολογία 35 προφορική άρχεται η ψηφοφορία πέρας ωραία επειδή έχει συνένα το ΕΛΚΑ ναι Συν ένα ΕΛΚ λοιπόν εγκρίνεται 36 άρχεται πέρας εγκρίνεται 5 5 άρχεται πέρας εγκρίνεται 39 άρχεται Πέρας. Εγκρίνεται. 41 άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. Εντάξει. 42 άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. 45 άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. 46 άρχεται. Πέρας. εγκρίνεται 47 άρχεται πέρας εγκρίνεται 48 άρχεται πέρας απορρίπτεται 50 άρχεται πέρας απορρίπτεται 51 άρχεται πέρας απορρίπτεται 52 άρχεται πέρας απορρίπτεται 53 άρχεται πέρας απορρίπτεται 54 άρχεται πέρας απορρίπτεται 55 άρχεται πέρας εγκρίνεται 56 άρχεται συγγνώμη συγγνώμη όχι συγγνώμη 58 πρώτα 58 άρχεται «58» λέω. Εντάξει. Πέρας. Απορρίπτεται. 56 άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. 57 άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. 59 προφορική άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. 60 άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. 61 άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. 62. Άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. 64 και 67 από κοινού. Πέρας. Εγκρίνονται. 66 άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. 68 άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. 71. Άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. Αιτιολογικές αναφορές 1. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται και αιτιολογική αναφορά, τροπολογία 2, άρχεται. <clears throat> Πέρας. Εγκρίνεται. Αιτιολογικές σκέψεις, τροπολογία 3, άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 4, άρχεται. Πέρας απορρίπτεται και το τελικό κείμενο, ονομαστική ψηφοφορία, άρχεται Ψηφίσατε όλοι. Όχι ακόμα. Πέρασε. εγκρίνεται 29 υπέρ 25 κατά μία αποχή Να προχωρήσουμε συνάδελφοι στην επόμενη ψηφοφορία Πρόταση απόφαση του Συμβουλίου για την εφαρμογή των διατάξεων του κεκτημένου του Σέγγεν στον τομέα συστημάτων πληροφοριών Σέγγεν στη Δημοκρατία της Κροατίας του κ. Μέλου. Μία ψηφοφορία, μέλο, ε, άρχεται ψηφοφορία. Πέραση της Εγκρίνεται. 50 υπέρ, 3 κατά, μία αποχή. Συγχαρητήρια στον κύριο Μέλλο. Επόμενο. Σχέδιο εκτελεστική απόφαση Συμβουλίου Αυτοματοποιημένη ανταλλαγή δακτυλοσκοπικών δεδομένων στη Λετωνία. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση ψηφοφορίας Εγκρίνεται. 47 ψήφοι υπέρ, 7 κατά, μία αποχή. Η συγκήτρια Τζούντιθ Τσαρτζεντίνη, αυτό με το οποίο είναι ανταλλαγή δεδομένων όσο αφορά τα δεδομένα DNA, άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση ψηφοφορίας. Εγκρίνεται 46 ψήφοι υπέρ, 6 κατά, 2 αποχές συγχαρητήρια. Τόμας Τζεντόφσκι, αυτομετωπιμένη ανταλλαγή δεδομένων όσον αφορά δακτυλοσκοπικά δεδομένα σε αρκετές χώρες. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 47 ψήφοι υπέρ, 6 κατά, 2 αποχές. Συγχαρητήρια στον εισηγητή. του αξίζει χειροκρότημα, θέλει και το χειροκρότημα. Θέλει και να μιλήσει, αλλά δεν θα του δώσω το λόγο. Κοσμενόβαστε συνέχεια, αντίστοιχο. Άδειε κυκλοφορία οχημάτων σε αρκετέ χώρε. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε τη ψηφοφορία. Εγκρίνεται 46 ψήφοι υπέρ, 6 κατά, 2 αποχές, συγχαρητήρια στην κυρία Χωισμόνεβα. Και τέλος, και κυκλοφορίας οχημάτων, ανταλλαγή δεδομένων σε αρκετές χώρες, Μαρία Γκραπίνη, άρχεται ψηφοφορία. Πέρασε της ψηφοφορίας. Συγχαρητήρια στην κυρία Γκραπίνη. Τέλος της ψηφοφορίας. Ευχαριστούμε τους συναδέλφους για την πειθαρχία τους. Σημείο 26 τώρα. Αν μπορείτε να αποχωρήσετε ησύχως, έχουμε και άλλους σημείο στην ημερήσια διάταξη. Έχουμε και άλλους σημείο στην ημερήσια διάταξη, δεν έχουμε επίτροπο. Σιλβί. Σιλβί. I'm so sorry. Ζητώ συγγνώμη. Ε, παραλογίζομαι. Στις δύο είναι το θέμα αυτό. Ζητώ συγγνώμη, Τζούντιθ. Συνάδελφοι, ζητώ συγγνώμη. Ε, μπορείτε να φύγετε για το γεύμα σας, να απολαύσετε και τη ζωή σας. Ο διάλογος για την ασφάλεια είναι στις δύο η ώρα. Σας παρακαλώ να είστε εδώ. Σας ευχαριστώ και ζητώ συγγνώμη. Καλή όρεξη. Κάτι άλλο σκεφτείτε.